Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Παρακαλώ να καθίσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν πιο ήσυχα. Θα ξεκινήσω με τις αποφάσεις των συντονιστών σήμερα το πρωί αιτήματα των ομάδων για ε, διαμόρφωση ημερησίων διατάξεων. Τον Απρίλιο θα δουλέψουμε πάνω στο Εθνικό Πάρκο Ντονάνα, στο πυρηνικό εργοστάσιο Γκαρόνα και στην αναφορά για την κύρωση της συνθήκης του Μαρακές. Όλα αυτά θα μπουν στη ημερησία διάταξη του Απριλίου για τη Λετωνία και την Εστονία και τα εκλογικά δικαιώματα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της δημόσιας ακρόασης για τους απάτριδες στις 29 Ιουνίου. Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών θα γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές και η ετήσια έκθεση για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή θα γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, οι συστάσεις που ήταν αντικείμενο διαφωνιών εγκρίθηκαν βάσει των δικών μου προτάσεων και κάποιες ε, αναφορές παραμένουν ανοιχτές για να δούμε τι θα γίνει με τη συνέχεια που θα δοθεί στα θέματα. Για τις διερευνητικές αποστολές και τις ακροάσεις αποφασίσαμε δύο διερευνητικές αποστολές να λάβουν χώρα στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 και κατά κύριο λόγο μία αποστολή θα γίνει στο Ταράντο, στην Ιταλία τον Ιούλιο και στη Λάρνακα της Κύπρου ε, τον Σεπτέμβριο και επικεφαλής αντιπροσωπείας για τη διερευνητική αποστολή στη Μαδρίτη αποφάσιστηκε να είναι η Τζουτ Κέρτεν Ντόλιν και το EFTD πρότεινε να γίνει μια κρόση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσωρινώς απασχολούμενων εργατών και θα γίνει αυτό το φθινόπωρο. Ε, στηρίξαμε το πρόγραμμα της ακρόσης για τη διάκριση σε βάρος ε, πολιτών στα κράτη-μέλη και την προστασία των μειονοτήτων. Η ακρόαση αυτή θα γίνει στις 4 Μαΐου και συζητήσαμε τη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής μας και αποφασίσαμε ενίοτε όταν τα ζητήματα είναι φλέγοντα και πιεστικά θα ενημερώνονται οι χρήστες μόνο στις γλώσσες που ε, αφορούν το κάθε θέμα. και μόλις είναι τεχνικός δυνατό, οι υποστηρικτές πίσω από τους, ε, τις αναφορές ε, θα λαμβάνουν ενημέρωση και κοινοποίηση για τη συνέχεια που έχει δοθεί στο θέμα τους και για το κατά πόσο έχουν ανέβει στην δικτυακή μας πλατφόρμα νέα καινούργια σχετικά έγγραφα και νέες σχετικές εξελίξεις. Εχθές ε, ξεκίνησε το γεγονός για το δίκτυο της Επιτροπής Αναφορών, την ε, Network. Είχαμε παριστάμενος από όλες τις ενδιαφερόμενες επιτροπές. Ήταν μια τεράστια επιτυχία που οργανώσαμε. Ας ελπίσουμε ότι οι συνάδελφοι θα παραμείνουν δεσμευμένοι και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτού του, αυτού του δικτύου. Συμφωνήθηκε επίσης να ε, μελετηθεί το ενδεχόμενο για σχέδιο διαχείρισης, διαχειριστικό σχέδιο για σαρκοφάγα ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ νοήτο μιλούμε για τους λύκου. Και μιλούμε και επίση στη συνέχεια για την συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες εγκρίθηκε και εγκρίθηκε και η τελική έκθεση για την ε, καλή διαβίωση των παιδιών, για την ευημερία των ε, παιδιών συμφωνήθηκε να υπερψηφιστούν οι τροπολογίες και το ΕΛΚ θα παρουσιάσει γνώμη έκθεση μειοψηφίας ίδιας πρωτοβουλίας. Δεν υπήρχε κάτι άλλο υπό τα διάφορα. Και αυτά έγιναν λοιπόν στη συνεδρίαση των συντονιστών. Τώρα ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Με χαρά σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με τους νέους διαδικαστικούς κανόνες που έχουμε εγκρίνει και που ισχύουν από 1η Πρώτου του 2017, προκειμένου να υπάρχει απαρτία στην Επιτροπή μας, πρέπει να είμαστε ε, ένα τρίτο παρόντα παρόν το 1 τρίτο των μελών. Άρα 12 βουλευτές πρέπει να είναι παρόντες για να υπάρχει απαρτία, άρα δικαιούμαστε να ψηφίσουμε και ψηφίσουμε την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας το 2015 τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8, α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 σε δύο τμήματα ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Όχι, συγγνώμη, καταπίπτει. Δεύτερο τμήμα δεν καταπίπτει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ.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 Όχι, λέει η Πρόεδρος. Καλώς. Το αποσύρουμε και ψηφίζουμε την τροπολογία 22. Ξεκινά η ψηφοφορία ηλεκτρονική για την τροπολογία 22. Πέρας της τροπολογίας. Και εγκρίνεται με μία ψήφο παραπάνω. Καλή, πολύ καλή προσπάθεια κύριε Πρέγκα. Δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 23 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. 26 την τροπολογία, 26 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 33, α, καταπίπτει, 33, 34, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36, υπέρ, κατά, αποχές, θα το ελέγξουμε, θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 36. Πέρες, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές θα το εγκρίνουμε ε, ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 38. Ξεκίνησε. Τώρα ξεκινάει, άνοιξε το σύστημα. Ψηφίζουμε την 38. Πέρας της ψηφοφορίας. Μακράν εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Η καλύτερη, κύριε Πρέντα, εγκρίνεται η καλύτερη τροπολογία. Τροπολογία 40 σε δύο τμήματα. Το πρώτο καταπίπτει. Και το δεύτερο παραμένει. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Επίσης καταπίπτει. Η τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σχέδιο γνωμοδότησης ως έχει. Έτσι όπως διαμορφώθηκε. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης μετά την ε, ψήφιση των τροπολογιών. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται σε μεγάλο βαθμό. Με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ θερμά. Και όσοι θέλετε να φύγετε από την αίθουσα μετά το πέρας της ψηφοφορίας, σας παρακαλούμε να το πράξετε γρήγορα και ησύχως. And now... Και τώρα ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο υπαριθμών 11 στην ημερήσια διάταξή μας. Πρόκειται για σημαντική συζήτηση. Πρόκειται για την τελική έκθεση της ομάδας εργασίας για θέματα παιδικής πρόνοιας. Θα εκτιμούσα οι συνάδελφοι να είναι ίσχυοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξή μας. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω τον λόγο. Καταρχάς, στην πρόεδρο της ομάδας εργασίας, κυρία Εύη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο έκθεση είναι το αποτέλεσμα των εργασιών μας ε, εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Εγώ είμαι πρόεδρος ε, της ομάδας εργασίας αυτής και σας παρουσιάζουμε σήμερα τα αποτελέσματα τέθηκαν διάφορα θέματα από αναφέροντες και θεωρήσαμε ότι κάποια από αυτά έπρεπε να εξεταστούν περισσότερο εις βάθος. Αν κοιτάξετε την εντολή μας, η ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με τέσσερις συγκεκριμένους τομείς. Εξετάσαμε λοιπόν θέματα με διασυνοριακές επεκτάσεις που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τέσσερις τομείς που εξετάσαμε είναι οι διασυνοριακές ε, απαγωγές ε, ανηλίκων από, από τους γονείς τους, ε, οι υπηρεσίες Jugendamt στη Γερμανία, οι υιοθεσίε χωρίς συγκατάσταση των γονέων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα εξαφανιστέντα βρέφη στην Ισπανία. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να εξετάσουμε και ένα πέμπτο θέμα, τις κοινωνικές υπηρεσίες στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οι αναλυτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν και με επαφές ε, με τους ε, αναφέροντες ε, ενδιαφερόμενους εμπειρογνώμονες και ε, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάσαμε στοιχεία, στατιστικές, ε, εθνικά μέτρα που θεωρήθηκε ότι, ε, δεν, ότι παραβιάζουν τον κοινοτικό νόμο. Εξετάσαμε επίσης το, την ομολογία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, είχα στη διάθεσή μου περιορισμένο προϋπολογισμό Κάλεσα όλες τις πολιτικές ομάδες να ορίσουν ε, εμπειρογνώμονες ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα ευαίσθητα για τις πολιτικές ομάδες θέματα. Σε περιπτώσεις που δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, εργαστήκαμε με τρόπο δημοκρατικό, ακολουθήσαμε την πλειοψηφία. Αυτά όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες που προσκλήθηκαν. Είχαμε πρώτα 8 συναντήσεις ε, όσον αφορά το αντικειμενικό περιγραφικό τμήμα της έκθεσης. Εκπονήθηκαν συστάσεις οι οποίες ε, μπορούν να τροποποιηθούν με τροπολογίες από όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού αποτελεί αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας εργασίας. Εξετάσαμε εξαντλητικά τα διάφορα θέματα, κάναμε πάρα πολλή δουλειά και προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όλα τα σημαντικά έγγραφα ε, ως παραρτήματα στο έγγραφο εργασίας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα έγγραφα θα είναι χρήσιμα για τους ε, όταν θα θέλουν να υποβάλουν τροπολογίες. Όσον αφορά τις ε, τελικές ε, συστάσεις που βρίσκονται στο τέλος του εγγράφου, τονίζουν την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κάτι που θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση και της νομοθεσίας. Ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους ανηλίκους. Έχουμε το συμφέρον του παιδιού κατά νου. Η, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν καθήκον να εξετάσουν και να αναλύσουν τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη-μέλη και που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις διαφορών για το δικαίωμα κυδαιμονίας ή επαφής με το παιδί. Πρόκειται για αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την, το παιδί. Υπάρχουν όμως κάποιοι τομείς όπου χρειάζονται περαιτέρω έρευνες. Με στόχο την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις ε, κακών πρακτικών. Ε, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, διότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, η ανταπόκριση που λάβαμε από τα κράτη-μέλη ήταν πολύ περιορισμένη. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις ε, για τα δικαιώματα των εμπλεκομένων. Θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να ε, διευκρινιστούν τα θέματα αυτά. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελιονόρα. Πράγματι ήταν ένα μακρύ αλλά σημαντικό ταξίδι. Σε ευχαριστούμε για όλη τη δουλειά που έχεις κάνει. Η ομάδα εργασίας έτσι ολοκληρώνει τις εργασίες της και παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσης. Το έγγραφο αυτό είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο ε, αναφέρει το αποτέλεσμα των διαφόρων συναντήσεων και το δεύτερο τμήμα είναι ο κατάλογος ε, συστάσεων. Στις συστάσεις μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες. Ε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 30 Μαρτίου στις 3 η ώρα. 30 Μαρτίου στις 3 η ώρα είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για τις συστάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τους συναδέρφους ε, να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Έχω πρώτο στον κατάλογο τον κύριο Βίλαντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου. Μη σας πω τον θυμό μου για τον τρόπο που αναφέρονται τα περί των υπηρεσιών νεολαίας στη Γερμανία, στο σημείο 4 του Jugendamt. Ανα Ε, αναφέρεται ότι πρόκειται για μια περίπτωση μιας ε, δημοσιογράφου κλπ. Πρόκειται όμως ε, και για ένα άτομο που έχει καταδικαστεί για που έχει καταδικαστεί για κάτι, οπότε με εκπλήσει ο τρόπος που εργάστηκε η ομάδα εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς που θα ήθελα να πάρει το λόγο από το S&D. Ο εκπρόσωπος του ECR, ο κύριος Μαριάς, δεν είναι παρόν. Α, Ρίκε, είσαι εδώ. Θέλεις να πάρεις το λόγο για το θέμα αυτό, όχι. Ούτε από την ΚΟΕ έχουμε κανέναν, ούτε από τους Πρασίνους. Εκτός μικροφώνου δεν ακούμε. Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό, ο Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε κουραστεί. Δεν πρόκειται για την πρώτη ομάδα εργασίας ε, που είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, είχαμε και αυτήν για την ε, Ισπανική Ακτοφυλακή και ήταν πολύ επιτυχής η εργασία της ομάδας αυτής. Είδαμε αποτελέσματα που οδήγησαν και σε τροποποίηση της νομοθεσίας στην Ισπανία. Η ομάδα εργασίας εργάστηκε με συνενετική διαδικασία και εργάστηκε με επιτυχία η ομάδα εργασίας αυτή. Ε, τούτη η ομάδα εργασίας ε, φαίνεται ότι δεν έχει εργαστεί με την ίδια επιτυχία. Ε, ε, εμάς το ΕΛΚ, η, εμάς το ΕΛΚ μας ενοχλεί στην ομάδα αυτή ότι δεν επιτεύχθηκε τελικά συνένεση. Έχουμε την εντύπωση ότι και διάφορες πολιτικές ομάδες ε, δεν ε, συμμετείχαν πολύ ενεργά και οι πληροφορίες ε, έφταναν αρκετά αργά σε εμάς. Όπως είπε και ο κύριος Βίλαντ όσον αφορά την κυρία Κολόμπο, βρίσκω ατυχές το ότι έχουμε μια αναφέρουσα η οποία ουσιαστικά αναφέρεται ως εμπειρογνώμων. Στην ε, έκθεση αυτή αναφέρονται οι ισχυρισμοί της κυρίας Κολόμπο χωρίς να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ισχυρισμούς ε, μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί στη Γερμανία. Επίσης, δεν ε, φαίνεται να έχει υπάρξει κάποιο συστηματικό λάθος, κάποια συστηματική κακή πρακτική στην ε, Γερμανία. Ο κύριος Χόφμαν είναι εκπρόσωπος ε, του Jugendamt, των υπηρεσιών νεολαίας, και θα μπορούσε να μιλήσει στην Επιτροπή μας. Ε, αντίθετα με την ε, κυρία Κολόμπο που είναι άτομο που έχει καταδικαστεί, ο κύριος Χόφμαν ε, θα μπορούσε να μας παρουσιάσει κάποιες απόψεις, αλλά αναφέρεται τελείως πανεπιπτόντος στο τέλος το όνομά του. Άλλωστε όλα αυτά εδώ πέρα είναι ισχυρισμοί της αναφέρουσας. Αυτό όμως θα έπρεπε να αναφέρεται σαφώς. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι με την ε, τελική έκθεση αυτή. Δεν πιστεύουμε ότι είναι μια έκθεση που βοηθάει την Επιτροπή Αναφορών. Το μόνο καλό είναι ότι ξανανοίγει έτσι η αναφορά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να κλείσει κιόλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κάρλσον. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, τελικά θα ζητήσω το λόγο. Έχω απόλυτο σεβασμό για τους Γερμανούς συναδέλφους που έχουν κάποιες επικρίσεις για το θέμα αυτό που επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας. Και φυσικά είναι απόλυτα θεμητό το να ε, σχολιάζει κανείς το πόσο έγκυρες είναι οι πηγές μας. Λυπάμαι όμως που τελικά ε, εκεί επικεντρώνεται η προσοχή, διότι νομίζω ότι όσο καιρό βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο, αυτή η εργασία είναι η πιο σημαντική που έχω κάνει. Ως πολιτικός, επί πολλά χρόνια έχω ασχοληθεί με κοινωνικές υποθέσεις, ιδιαίτερα υποθέσεις που αφορούν παιδιά. Και στην ομάδα εργασίας αυτήν, πέρα από το ότι πιθανότατα να υπήρχαν διαφορετικοί ε, λόγοι για την ύπαρξη αυτής της, πολιτικής, ε, αυτής της ομάδας εργασίας, ε, θα συμφωνήσω με την Ελεονόρα Εύη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που μπορέσαμε να ασχοληθούμε με υποθέσεις από όλη την Ευρώπη και πιστεύω ότι ήταν σημαντικό για την ομάδα εργασίας να διαπιστώσει ποιοι είναι οι συνδετικοί κρίκοι, ε, ποια είναι η γενική κατάσταση για τα παιδιά στις περιπτώσεις όπου πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους οι διάφορες χώρες. Επίσης, ε, πιστεύω ότι ε, είναι αρκετά δύσκολο να μας επικρίνει κανείς τη στιγμή που δεν είχαμε περισσότερους πόρους. Εγώ θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να εξετάσουμε περισσότερες υποθέσεις. Είχαμε διάφορες ενδιαφέρουσες συζητήσεις που νομίζω ότι θα μπορέσουν να είναι σημαντικές και για τις εργασίες μας εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, και κατά την επιλογή των ε, θεμάτων ε, με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε από νομοθετικής πλευράς ε, και θέλουμε να υποβάλουμε συστάσεις για το μέλλον. Με όρο το σεβασμό για τα όσα είπατε και βέβαια πάντα πρέπει να προσέχουμε ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των επιρογνωμόνων μας, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά καλά που θα μπορούσε να πει κανείς για τη δουλειά που έγινε σε αυτή την ομάδα εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ροζιέρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα καλά το πρόβλημα. Είμαι νέα σε αυτή την Επιτροπή και τώρα καταλαβαίνω τον τρόπο λειτουργίας, όμως το πρώτο μέρος αναφέρεται στο πρόβλημα που είναι η αποκατάσταση των λόγων των εμπειρογνωμόνων που προσκλήθηκαν. Αυτό δεν δεσμεύει την ομάδα. Ποια θα ήταν η αναλλακτική από ό,τι καταλαβαίνω ασκείται κριτική στα λόγια των εμπειρογνωμόνων ή στην ικανότητά τους. Αλλά από τη στιγμή που τους προσκαλέσαμε ως εμπειρογνώμονες και ειδικού και τους ζητήσαμε να πάρουν το λόγο με αυτή την ιδιότητα, φυσικό μου φαίνεται να τους αποδώσουμε τα λόγια τους. Βεβαίως που θα γίνουν αντικείμενο συζήτησης, αλλά πώς ε, θα μεταμφιέσουμε ή θα λογοκρίνουμε ή θα τροποποιήσουμε λόγια που δήλωσαν και που είπαν ως εμπειρογνώμονες όταν εμείς τους καλέσαμε ως τέτοιου, δεν μου φαίνεται αυτό δυνατό να γίνει. Θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα ποια ήταν τα λόγια των εμπειρογνωμόνων και ποια είναι η γνώμη που θα υιοθετήσει η Επιτροπή. Ομολογώ ότι εκπλήσωμαι, προβληματίζομαι. η δουλειά που έγινε έχει συνέπεια και είναι αρκετά ολοκληρωμένη, άρα είναι απαραίτητο να αποδώσουμε στους εμπειρογνώμονες ε, ε, τις δηλώσεις τους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βίλαντ έχει το λόγο για σύντομη παρέμβαση. Χαίρομαι που στο μεταξύ συμφωνήσαμε σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να εργάζεται η Επιτροπή μας όσον αφορά τις διερευνητικές εργασίες και τις ομάδες εργασίας. Γι' αυτό δεν θα υποβάλω τροπολογία. Έχει καταγραφεί το τι έγινε στην ομάδα εργασίας και η κυρία Ροζιέρα έχει απόλυτα δίκιο. Δεν ε, έχω επικρίνει το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό. αυτό. Αυτό που ε, επικρίνω ε, είναι η επιλογή των ε, εμπειρογνωμόνων. Κυρία Άουκεν, συγγνώμη, μου επιτρέπετε να τα λέω αυτά. Εκτός μικροφώνου παρατήρηση. Κυρία Άουκεν, συζητάμε την έκθεση αυτή και είναι δικαίωμα της Επιτροπής μας να ε, λέμε τη γνώμη μας. Το δικαίωμα αυτό το ε, ασκείτε και εσείς ε, πολύ συχνά σε περιπτώσεις διαφόρων εκθέσεων. Θα ήθελα να πω ότι δεν θεωρώ την κυρία Κολόμπο εμπειρογνώμονα, την θεωρώ ενδιαφερομένη. Ανέφερα και κάποια άλλα επίθετα τα οποία δεν θα επαναλάβω, αλλά είναι ένα άτομο με μία άποψη, μία ενδιαφερομένη. Σε τέτοια περίπτωση λοιπόν, ε, η ισορροπία δεν είναι πολύ καλή, διότι ε, το μεγαλύτερο τμήμα ε, του τμήματος αυτού της έκθεσης αναφέρεται στη δική της γνώμη, ενώ για τους άλλους δίνονται πολύ λιγότερος χώρος. Και κυρία Όκεν, ναι, έχω δικαίωμα να σου το δικαίωμα αυτό. Το δικαίωμά μου το λόγο. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο. Όμως, ζητώ από τους συναδέλφους, όταν συνεδριάζει η Επιτροπή μας, να μην κάνουν μορφασμούς την ώρα που μιλάει ο άλλος, να προσπαθήσουν να είναι όσο να πιο ευγενείς. Αυτό θα διευκολύνει τη ζωή όλων μας. Και ε, θα δώσει και καλύτερη εντύπωση για το θεσμικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Επιτροπή των Αναφορών. Θα δώσει καλύτερη εικόνα στους αναφέροντες, στους πολίτες της Ευρώπης, οι οποίοι τα παρακολουθούν όλα αυτά. Μεταδίδεται διαδικτυακά η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Παρακαλώ. Μάργαρετ, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία ε, Δασκάλα. Να πω ότι μερικές φορές μέχρι και το ΕΛΚ φτάνει αργά Όλα αυτά έχουν γίνει, είναι περασμένα, είναι έτοιμα και γι' αυτό είναι τόσο φορτωμένο το πρόγραμμα στην Επιτροπή μας. Γιατί καθόμαστε και συζητάμε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι περασμένο, ξεχασμένο, κάτι το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει ήδη γίνει. Εκτός μικροφώνου οι ομιλητές, η πρόεδρος Μπορεί κανεί να συμφωνήσει με αυτό που λέτε ή να διαφωνήσει. Εγώ έχω τη δική μου θέση και τη γνωρίζετε οι περισσότεροι. δεν είναι η μόνη εμπειρογνώμονα η κυρία Κολόμπο και άλλοι εμπειρογνώμονες στο κείμενο ε, αναφέρονται και λέμε σύμφωνα με τον τάδε και τάδε και τάδε αυτό είναι το πλαίσιο. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει ε, στο τμήμα των συστάσεων γιατί αυτό θα αντικατοπτρίσει τη θέση της Επιτροπής μας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σέιβη και θα κλείσω τον κατάλογο μιλητών για το θέμα αυτό κάπου εδώ και θα δώσω μετά το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, η Ελεονόρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Καταρχάς, ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων διαμορφώνεται ε, κατόπιν δημοκρατικής διαδικασίας γιατί έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας της Επιτροπής. Και αυτό συμβαίνει με όλες ε, τις ακροάσεις και τους εμπειρογνώμενες και ειδικού που έχουμε καλέσει στις εκάστοτε ομάδες εργασίας μας. Οφείλω να το πω και λυπούμε που το λέω, ε, οφείλω να πω το εξή. Ε, Κάποιε ομάδε, ειδικά το ΕΛΚ, πότε δεν παρουσίασαν κανέναν εμπειρογνώμονα και πολύ συχνά άσκησαν κριτική στη συγκεκριμένη εμπειρογνώμονα για το Jugendamt, αυτό το ε, ε, ταμείο για τα παιδιά ε, στη Γερμανία, ή Άλλες φορές για άλλους εμπειρογνώμονες το ΕΛΚ έχει εκφραστεί προκλητικά ε, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια των ε, προσκεκλημένων μας και λείπουμε πολύ που οφείλω να το πω αυτό εδώ δημόσια και το λέω. Θέλω επίσης να διευκρινίσω ότι στο τελικό κείμενο ε, βάλαμε ένα disclaimer, ένα, μια ειδοποίηση, γνωστοποίηση, υποσημείωση, όπως θέλετε πείτε το, όπου δηλώναμε ότι οι, οι, θέσεις των ε, εμπειρογνωμόνων εκφράζουν τους ιδίους και σε ουδόλως εκφράζουν τη θέση της ε, Επιτροπής μας. Επομένως, οι επισκέψεις επιτόπου στο παρελθόν, η η παρέμβαση της εκπροσώπου του Jugendamt στην Επιτροπή των Αναφορών κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών. Όλα αυτά είναι στοιχεία που δεν έχουμε εξετάσει κατά τη διάρκεια των συσκέψεων της ομάδας εργασίας και των ομάδων εργασίας. Άρα δεν έχει κανένα νόημα, κατά τη γνώμη μας, να τα αναφέρουμε όλα αυτά στο περιγραφικό σκέλος του τελικού εγγράφου. Αλλά παρόλα αυτά, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα ορισμένων πολιτικών ομάδων, αποφασίσαμε να έχουμε ένα παράρτημα αυτών των στοιχείων των ενημερωτικών στο τελικό έγγραφο για λόγους ενημέρωσης χωρίς καμία περαιτέρω ε, πολιτική ερμηνεία για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται στην εκάστοτε αποστολή. Επομένως, επαναλαμβάνω ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ε, βασίστηκε σε μεγάλη δημοκρατική και διάφανη συμμετοχή. Και με τον τρόπο αυτό και δια της πλειοψηφίας ελήφθησαν οι αποφάσεις. Thank you very much. Now, the Commission representative... Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία του το παρακαλώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Thank, thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει γνώση και θα ε, τη λάβουμε υπόψη κατά τις εργασίες μας για τα δικαιώματα του παιδιού. Ε, αναφέρεται βέβαια περισσότερο ε, στα δικαιώματα των γονέων παρά των ε, δικαιωμάτων του παιδιού. Αναφέρεται περισσότερο στο δικαίωμα κυδαιμονίας. Θα ήταν χρήσιμο η έκθεση να παραπέμπει στα διεθνή πρότυπα που διέπουν τον τομέα αυτών. Για παράδειγμα, η Γενική Παρατήρηση, ε, σημείο 14, της, ε, ιδιαίτερα το τμήμα 5β, ε, σχετικά με τα διαδικαστικά εχέγγυα της ε, Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού διότι τα διαδικαστικά εχέγγυα που συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ καλά και όλα θα ήταν καλύτερα εάν όλοι τα εφαρμόζαμε. Επίσης, ε, γενική παρατήρηση υπαριθμών 14. Γενική παρατήρηση 13 σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού για ε, ελευθερία από κάθε μορφή βίας. Ε, μπορεί να αφαιρεθεί από τους γονείς το παιδί σε περίπτωση που ε, ασκείται βία ή που ε, ε, υφίσταται σημαντικές στερήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή θεωρείται απαραίτητο να απομακρυνθεί το παιδί από την κυδαιμονία των γονέων και εξετάζεται η αναλογικότητα και η καταλληλότητα των μέτρων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ χρήσιμη η αρχή αυτή. Οι 10 γενικές αρχές για τα σχετικά συστήματα αναφέρονται στο πρώτο τμήμα της έκθεσης. Ε, το Κοινοβούλιο όμως ε, θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει να εφαρμοστούν. Αναγνωρίζεται η οικογένεια ως ε, ο πρώτος παράγοντας φροντίδας και θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην οικοδόμηση δυναμικού στον τομέα της ε, προστασίας ε, των παιδιών. Επίσης, ε, η φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Όσον αφορά την αρχή του κατεπήγοντος για όλες τις διαδικασίες όπου συμπεριλαμβάνονται παιδιά, θα πρέπει να αναγνωριστεί και αυτή η αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Εύη, θέλετε να απαντήσετε στα όσα υπόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, ωραία. Ωραία. Ξανατονίζω λοιπόν την σημασία να ξανακοιτάξετε τις συστάσεις στο σχέδιο έκθεσης και να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας πριν τις 3 το απόγευμα στις 30 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ και προχωράμε στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο 12. Ε, πολύ καλά προχωράμε. Είμαστε ε, μπροστά στο πρόγραμμα. Ε, δεν είναι εδώ οι αναφέροντες ακόμα, είναι εδώ όμως εκπρόσωπος της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά υπαριθμών 1134-2015 ε, σχετικά με την οργάνωση της εργασίας στα πλοία από ναυτιλιακή εταιρεία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο κατευθείαν στην κυρία Καρθία Καρθία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή, καλό απόγευμα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απήντησε ήδη γραπτά ε, εις τον ε, αναφέροντα στις 3 ε, Αυγούστου του 2016 και ότι στην απάντησή μας λέγαμε ότι μια και πρόκειται για ιδιαίτερη κατάσταση, δεν μπορούμε να ε, συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα, κυρίως γιατί αφορά ένα ιταλικό θέμα, δηλαδή συνθήκες εργασίας σε ένα ιταλικό πορθμίο. Ε, οι διοικητικές και δικαστικές αρχές είναι, της Ιταλίας είναι αυτές οι οποίες ε, έχουν και υπό το φως του ευρωπαϊκού δικαίου την ε, αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να ελέγχουν τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. το προηγούμενο μήνα λάβαμε συμπληρωματικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να μεταφραστούν ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα εξετάσουμε. Έχουμε ήδη μεταφράσει ορισμένα. Ε, τα κείμενα τα οποία διαβάσαμε μετά από τη μετάφρασή τους ε, δεν τροποποιούν την αρχική μας τοποθέτηση, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μετάφραση όλων των εγγράφων ε, και τότε θα μπορέσουμε να δώσουμε την γραπτή μας απάντηση. Θα την αποστείλουμε στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Οι συνάδελφοι, παρακαλώ, έχουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις. Απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οφείλω να πω και να ομολογήσω ότι αν δεν είχατε πει ότι παραμένουν κάποιες μεταφράσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα και έτσι θα διευκρινιστούν διάφορες λεπτομέρειες. Η κατάσταση μέχρι τη δήλωσή σας ήταν πια ότι η αξιολόγηση της κατάστασης καθιστά σαφές ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ενσωματώσουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες στην εθνική τους νομοθεσία. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου φέτος, άρα περίπου έχουμε ένα εξάμεινο αναμονής. Όμως το συγκείμενο καθιστά σαφές ότι είναι ευθύνη των εθνικών αρχών. Άρα κατανοώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει καμία επιλογή να δράσει. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Όμως, γνωρίζοντας την Επιτροπή, τους ανθρώπους ονομαστικά τους, ε, αρμοδίους, στην αντίστοιχη γενική διεύθυνση, θεωρούν ότι η δουλειά τους δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα, παρακολουθούμε και εμείς τα ε, πεπραγμένα της Επιτροπής και περιμένουμε να μας κάνετε τις τελικές δηλώσεις. Ευχαριστώ. Η Ελεονόρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και έτσι ώστε να μεταφραστούν όλες οι συμβληματικές πληροφορίες και να αξιολογηθούν σωστά, αλλά και για κάποιο άλλο λόγο. Προτείνω να στείλουμε επιστολές ενδεχομένως εις τον ε, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών, αλλά και στην επιθεώρηση εργασίας της Ενάπολης, έτσι ώστε να ε, ρωτήσουμε, να ζητήσουμε ε, τον έλεγχο της ε, σωστής εφαρμογής των κανόνων, γιατί παραμένουν πολλές φεζόνες. τα στοιχεία τα οποία αναφέρουν οι αναφέροντες και που καταγράφονται στην, αναφορά τους είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά και επομένως νομίζω ότι για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Κύριε Μπέκερ. Έχουμε χρόνο. Πέστε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο ομιλήτρια προηγουμένως, η συνάδελφος, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Αλλά μη λησμονήσετε όταν θα πάτε την τελική σας απόφαση ότι ε, θα πρέπει να μας ε, πείτε ακριβώς ε, τι έχει γίνει και, εν πάση περιπτώσει, να κινητροδοτήσουμε τον αναφέροντα ε, να ε, ξέρει τι να κάνει, για, αν θα πρέπει να ε, πάει στα εθνικά δικαστήρια για να βρει το δίκαιο του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κρατάμε το θέμα ανοιχτό μέχρι ότου ολοκληρωθεί η εξέταση από βάση Κομισιόν των Συμπληρωματικών Στοιχείων και όταν θα αναλυθούν όλα αυτά θα μας θα κοινοποιήσετε την απόφασή σας. Εν τω μεταξύ όμως θα στείλουμε και τις επιστολές στην Ιταλία ε, επιμένοντας και επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να εφαρμόζονται να, σωστά ε, οι ε, οδηγίες και τα νομιωτικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, να στείλουμε και μία επιστολή και στον αναφέροντα, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς έγινε, λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά του 2015, να του πούμε ακριβώς τι έχει γίνει και ότι εν πάση περιπτώσει ε, να του ε, πούμε ότι οι ε, αρχές θαλασσίου, η επιθεώρηση εργασίας, οι αρχές ελέγχου θαλασσίων υποθέσεων και τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διατάξεως είναι πολλά τα θέματα. Είναι τα σημεία 13, 14, 14, 15 και 16 ε, στη, της Διατάξεως έχουμε εδώ τους αναφέροντες εξαίρετα, άψογα, υπέροχα και συνεχίζουμε. Ε, παρακαλώ, ε, θα, θα περιοριστείτε σε τρία λεπτά ο καθένας γιατί είστε πολλοί. Πρώτα απ' όλα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πιέρ Παόλο Βόλπε και μετά την κυρία Ελίζα Ντιματέα. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Πιερ Πάολο Βόλπε, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, επιτρέψτε μου, ε, ε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ε, δυνατότητα να καταγγείλω και ενώπιόν σας για μία ακόμα φορά τις, τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι Ιταλοί συμβασιούχοι. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τόσο καταχρηστικά οι συμβάσεις ορισμένου ε, ακόμα και ο Άριος Πάγος της ε, Ιταλίας ε, πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις λέγοντας ότι είναι αντισυνταγματικές αυτές οι διαρκείς ανανεώσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, ειδικά στην επαρχία της Απουλίας ήταν πάνω από 2.000 οι εργαζόμενοι με τέτοιου είδους συμβάσεις. Μιλάμε για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που όμως έχουν πίσω τους οικογένειες οι οποίοι δεν μπορούν ε, να δώσουν αξιοπρεπή ζωή στα παιδιά τους, δεν μπορούν να οραματιστούν το μέλλον με τις οικογένειές τους. Γι' αυτό λοιπόν το Ιταλικό κράτος θα πρέπει οπωσδήποτε και άμεσα να σταματήσει αυτές τις συμβάσεις αυτού του είδους και θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, μην επιτρέψει την ανανέωση για τους συμβασιούχου που έχουν ξεπεράσει του 36 μήνε. Η πρόεδρο λέει παρακαλώ πολύ μιλάτε με τρομερά μεγάλη ταχύτητα, οι διερμηνεί δεν μπορούν να σα ακολουθήσουν. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε από το Ιταλικό κράτο, να θυμίσουμε στο Ιταλικό κράτο και την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ε, κάθε μέρα που περνάει με τέτοιου είδους ε, συμβάσεις σημαίνει ότι ζημιώνονται με τον χειρότερο τρόπο και καταπατώνται τα δικαιώματα των εργαζομένων και βεβαίω θα πρέπει ε, να ε, συνεχιστεί, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση τη στιγμή μάλιστα που ήδη υπάρχει απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου που λέει ότι όταν ξεπεραστούν οι 36 μήνε, τότε πρέπει οπωσδήποτε η σύμβαση ορισμένου χρόνου να μετατραπεί και να γίνει αορίστου χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να σας πω ότι ήδη στις 22 ε, Δεκεμβρίου του 2016 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, έστειλε επιστολή σε την αρμόδια Ιταλική Αρχή για ενδεχόμενη παραβίαση νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα δεν έχει γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκώς μας υπόσχεται, αλλά οι υποσχέσεις μένουν κενό γράμμα και τελικά δεν λύνεται το πρόβλημα αυτής ε, της ασάφειας. Ε, για μία ακόμα φορά λοιπόν οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ε, βρίσκονται σε μία κατάσταση δύσκολη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβάσεις πολλών ε, νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να απαιτήσει από, την Ιταλική, από τις Ιταλικές αρχές να λύσει για, μία, ε, ε, τελειωτικά συγγνώμη, και τελεσίδικα αυτό το πρόβλημα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που διαρκώς ανανεώνονται. Σας ευχαριστώ πολύ much Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξεπεράσατε το χρόνο σας. η κυρία Ελίζα Ντι Ματέο, η οποία ε, εκπροσωπεί τον κύριο Μπαρναμπά. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Εγώ είμαι η δικηγόρος ε, του ε, κυρίου Ντάβιντε Μπαρναμπά και μιλώ εξ ονόματός του. Ε, ο κύριος Μπαρναμπά λοιπόν το 25 Μαΐου του 2001 προσελήφθη από την περιφέρεια της Σικελίας ε, με, μια σύμβαση ορισμένου χρόνου. 19 φορές λοιπόν παρατάθηκε, ανανεώθηκε αυτή η σύμβαση για 15 χρόνια. Ε, ακριβώς για τον λόγο αυτό ο, ε, και επειδή μάλλον το, η σύμβασή του δεν έγινε ε, αορίστου χρόνου, ο αναφερόμενος αναγκάστηκε να στραφεί προς το δικαστήριο της ε, Κατάνια το τμήμα εργασιακών θεμάτων, αλλά η πρώτη ακρόαση έχει προβλεφθεί για την 22η Πρώτου του 2019. Καταλαβαίνετε ότι ε, παρότι ο, ο άνθρωπος αυτός έχει ε, εδώ και 15 χρόνια εργαστεί για το καλό της πόλης, δεν έχει ανανεωθεί, δεν έχει τροποποιηθεί ενισχυθεί η σύμβασή του έτσι ώστε να γίνει ορισμένου χρόνου. Ε, άλλωστε, η ίδια η επιθεώρηση εργασίας αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 36 ε, του νόμου 2001 του ε, υπαριθμών 165, ούτως ή άλλως αυτή η παροχή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και επομένως θα πρέπει να καταδικαστεί η περιφέρεια. Επίσης, το ε, επίσης να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν παρόμοιες ε, αποφάσεις ε, από προηγούμενα χρόνια. Όμως φαίνεται ότι η νομολογία δεν δίνει την δυνατότητα για αποζημίωση και παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί σε μια κατάσταση όπου υφίστανται την διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους τους οι οποίοι έχουν απεριορίστου χρόνου ε, και καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες. Ε, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η περιφέρεια της Σικελίας ε, παραβιάζει και τις, τους Ιταλικούς νόμους αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα ε, με τη μη διακριτική μεταχείριση. Επίσης, το άρθρο 13, εδάφιο 2 του νόμου 165 του 2001 αναφέρει σαφώς ότι ε, θα πρέπει οπωσδήποτε μετά από συγκεκριμένες παρατάσεις οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου να, στραφούν, ε, να μετατραπούν μάλλον σε αορίστου χρόνου εκτός και αν προκύπτουν ε, συγκεκριμένες συνθήκες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ε, Γι' αυτό λοιπόν ε, ζητούμε από, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μια διαδικασία επιπαραβάση έναντι της, ε, ε, επί... της περιφέρειας της Σικελίας. Ο κύριος Μπαρναμπά ζητά γρήγορη ταχεία αντιμετώπιση του θέματος και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατέψει αυτούς τους εργαζόμενους και να καταδικάσει ή μάλλον να ανοίξει διαδικασία επιπαραβάση έναντι των υπευθύνων Αθήνων. Πρόεδρος, γνωρίζω ότι έχετε πολλά πράγματα να πείτε, προσπαθήστε όμως... A possible chance to, to interpret and make your information available to everybody. Now, the next... Προσπαθήστε πάντως να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί δεν θα είναι σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Ευχαριστώ. The petition number 400. Εκπροσωπεί την αναφορά 413. Παρακαλώ, η Κλάρα. Κιάρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Αντωνίνο. Ε, όπως και ο κύριος Μπαρναμπά ε, έχουν ε, τον Μάιο του, έχει το 2001 τον Μάιο ε, προσληφθεί από την ε, ε, περιφέρεια της Σικελίας. Για 15 χρόνια έχει το ίδιο αυτό συμβόλαιο, δηλαδή είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν ανανεωθεί 19 φορές. Ε, σε μερικές ε, περιπτώσεις ε, έχουν υπάρξει κάποιες διατάξεις οι οποίες, οι οποίες επιτρέπουν αυτήν την διαρκή ανανέωση ενώ η σύμβαση δεν θα έπρεπε να έχει ξαναανανεωθεί. Πρόκειται για εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ε, της ε, ε, περιφέρειας. Επί χρόνια λοιπόν ε, η ε, περιφέρεια έχει ε, καταπατήσει, έχει παραβιάσει και εθνικό δίκαιο και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως ζητούμε να υπάρξει παρέμβαση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι της περιφέρειας της Σικελίας η οποία εξακολουθεί να ακολουθεί την ίδια πρακτική της παράτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ο κύριος ε, Τροβάτο, ακριβώς επειδή προσπάθησε να βρει το δίκαιο του, ε, ήδη ε, πήγε στο δικαστήριο της Κατάνια, αλλά η πρώτη του ακρόαση έχει οριστεί για την 9η Ιουλίου του 2018. Είναι προφανές λοιπόν ότι μέχρι σήμερα ο κύριος Τροβάτο με κανένα τρόπο δεν έχει καλύψει τα δικαιώματά του που έχει ως εργαζόμενος, ούτε από άποψη νομοθετική, ούτε από άποψη σε της εργασίας του. Ε, ε, και ούτε βεβαίως έχει υπάρξει οποιοδήποτε ε, νομικό μέτρο μέχρι τώρα. Αυτές οι ατελείωτες παρατάσεις των συμβάντων των συμβάσεών του ε, οπωσδήποτε δεν συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Άλλωστε πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, συγκεκριμένα με την απόφαση της 26 Νοεμβρίου 2014 όπου αναφέρει ότι θα πρέπει σε περίπτωση που ε, καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες να υπάρξουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου διαφορετικά ε, παραβιάζεται το εδάφιο 5 του ε, σημείου 1 ε, γράμμα α της οδηγίας 1999 κάθετος 70 στην ε, ε, ουσία υπάρχουν κάποιες ε, ποινές οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ χαμηλές και επομένως δεν είναι αποτρεπτικές και οι αρχές της Σικελίας εξακολουθούν να, να ακολουθούν την ίδια πρακτική χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ούτε την βιολογική ούτε την υπαξιακή ζημία των εργαζομένων. Ε, Επομένω, και ο εργαζόμενος τον οποίο εγώ σήμερα εκπροσωπώ αλλά και οι εργαζόμενοι υπόλοιποι που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση ε, ζητούν να παρέμβετε για να σταματήσει η κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Μαρία Καρμέλα Αντιματέα είναι η επόμενη ομιλήτρια. εκπροσωπή του αναφέροντα της αναφοράς 0422. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρία Πρόεδρε, της Επιτροπής, ε, ε, εγώ λέγομαι Ντιματέα Μαρία Καρμέλα και εκπροσωπώ την κυρία Μαγκάνο Πάολα Ντανιέλα. Η κυρία Μάγκανο ε, είναι και αυτή ε, μια εργαζόμενη η οποία προσελήφθη από την Ερτζόνε Σιτσίλια στις ε, 25 Μαΐου του 2001 βάσει ενώ μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Εργάστηκε ε, ε, πάντα από το Μάιο μέχρι το 2001 μέχρι και τώρα ε, με τέτοιες συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονται. Οι, της, οι δικές της συμβάσεις έχουν ανανεωθεί 18 φορές. Πρόκειται για μία αρχιτεκτόνησα η οποία πάντοτε και με εξαιρετικό τρόπο έχει καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η κυρία Μάγκανο ε, ε, έχει ε, καλύπτει έκτακτες ανάγκες της περιφέρειας. Ήδη από το 2002 έχουν είχε εργαστεί σε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην Έτνα καθώς επίσης και ασχολήθηκε και με τον σεισμό στο Αμπρούτσο το 2009 και στην Εμίλια το 2012. Ε, είναι επομένως προφανές ότι η κυρία Μάγκανο όλα αυτά τα χρόνια ε, ήταν ε, υπάλληλο της δημόσιας διοίκησης πάντα με τις ίδιες υποχρεώσεις. Έχουν υποβληθεί πάρα πολλές ε, ε, προτάσεις ε, και από το Κοινοβούλιο της Σικελίας, αλλά παρέμειναν κενό γράμμα. Εστράφει λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Μάγκανο, στην επιθεώρηση εργασίας της Σικελίας. Ωστόσο, ε, και στην προκείμενη περίπτωση, ενώ έγινε αποδεκτό το αίτημά της προς ε, διερεύνηση, η πρώτη ακρόαση έχει οριστεί για την 23η Πρώτου του 2019. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν ζητούμε να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση έναντι της ε, περιφέρειας της Σικελίας, έτσι ώστε να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα αυτής της κυρίας. Ευχαριστώ Thank you Ευχαριστώ πολύ. Αλεσάνδρο Ντιφέντε, εκπροσωπώντας τους αναφέροντες στην αναφορά 0429. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ ε, που παρακολουθείτε το θέμα μας. Η κατάσταση της κυρίας ε, Ροσάντζολα Κονσεντίνο, την οποία εκπροσωπώ, είναι παρόμοια με, τους, ε, με τις άλλες περιπτώσεις που ήδη παρουσιάστηκαν. Το συμβόλαιο της αναφέρουσας έχει για μία ακόμα φορά και για δέκατη η φορά, λέω, ανανεωθεί. Εδώ και 15 χρόνια λοιπόν ε, εργάζεται εις την ε, ε, lo Stato, eppure ancora a loro vengono negati i diritti. Στην πολιτική προστασία καλύπτοντας συγκεκριμένες και παρόμοιες ανάγκες. Λαμβάνοντας υπόψη όμως την λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ε, ε, εδώ πρέπει να σημειώσω ότι αφενός υπάρχει παραβίαση, αφετέρου όμως η ζημία ενδεχομένως δεν θα αφορά μονάχα την ε, κυρία που είναι η αναφέρουσα, αλλά και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Να σας πω ότι, το, ότι η χωροθέτηση, η προστασία και η πρόληψη και η διαχείριση ανάλυση κινδύνων ε, από σεισμού ε, και από ηφαίστεια ε, σε μια περιφέρεια η οποία είναι ιδιαίτερο σεισμογενής και παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο όσον αφορά τα ηφαίστεια, διότι πρόκειται για ηφαιστειογενή ζώνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα θέματα, λέω, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από ανθρώπους που είναι βέβαιοι ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους αυτού του είδους ε, οι εργασίες δεν είναι δυνατόν να αφήνονται στα, στην τύχη από πλευράς της δημόσιας διοίκησης. Είναι πάρα πολύ σοβαρές θέσεις, είναι θέσεις ευθύνης και επομένως ε, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ε, ότι η Ιταλία παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλους κινδύνους. Επομένως, το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως ε, κάνουν καλά τη δουλειά τους, ε, ε, δεν μπορούν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο έτσι ώστε να δουλέψουν καλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι μονάχα για εκλογικούς λόγους δεν ανανεώνονται, δεν μετατρέπονται οι συμβάσεις αορίστου χρόνου, σε, συγγνώμη, ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου, καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητούμε να επιληφθείτε του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι επόμενες δύο αναφορές, οι επόμενοι δύο ομιλητές εκπροσωπεί ο καθένας από δύο αναφορές. Έχουμε τον Σέρτζιο Καλεάνο, το δικηγόρο που ε, εκπροσωπεί τον αναφέροντα 988 και 1011 του 2016. Από τη στιγμή που εκπροσωπείτε δύο αναφέροντες πρέπει να έχετε διπλάσιο χρόνο ομιλίας, θα έχετε έξι λεπτά μαζί με την παρουσίαση PowerPoint που έχετε να κάνετε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, και τους εκπροσώπους ε, της ε, Κομισιόν. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία υπόθηκαν ήδη και τα έχετε ακούσει. Ωστόσο πρέπει να υπενθυμίσω ότι ε, στην ε, ε, Ιταλική νομοθεσία προβλέπεται η τροποποίηση έτσι όπως αναφέρεται άλλωστε και στην απόφαση αφατάτο στην περίπτωση κατά την οποία δηλαδή η Ιταλική κυβέρνηση ζήτησε την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχουμε επίσης και την απόφαση Μάσκολο του 2000 2014 με αριθμό C22 ε, κάθετος 13 ε, και μάλιστα και στην Ιταλία ε, το συνταγματικό δικαστήριο βασιζόμενο και στην απόφαση μάσκολο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απεφάνθη ότι όντως υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης. Η Ιταλική νομοθεσία, κυρίως αυτή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ανωτότων Ερετικού ε, Δικαστηρίου ε, αναφέρει σαφώς ότι ε, υπάρχει αξίωση αποζημίωσης ωστόσο δεν λόγω του ότι έπρεπε να παραχθούν τα πιστήρια της ζημίας έτσι ώστε να προκύψει η αποζημίωση παρέμεινε η απόφαση αυτή κενό γράμμα μέχρι την απόφαση 368 κάθετος 2000 ε, σύμφωνα με την ε, τελευταία απόφαση ε, για την περίπτωση ας πούμε των εργαζομένων είτε στη Σικελία είτε εργαζόμενους στον τομέα της δημόσιας υγείας σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει η αποζημίωση από 2,5 μέχρι 12 μήνες. Έχουν υπάρξει και άλλες ε, πολύ αρνητικές παρεμβάσεις ε, ε, που αναφέρονται άλλωστε και στις στα γραπτά μας σχόλια, τα οποία στείλαμε σε εσά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα αναφέρω εδώ. Υπενθυμίζω και σε σχέση με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι από τη Σικελία ότι υπάρχουν καταστάσεις ακόμα χειρότερες από αυτήν ε, που έχουν αναφερθεί προηγουμένως. Ε, ε, υπάρχει μία απόφαση του εφεσιδικίου της Κατάνιας που αναφέρει ότι σε περιπτώσεις εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες ή διαρκείς ανάγκες δεν ε, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ε, ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία διότι ε, στην αρχή οι συμβάσεις αυτές δημιουργήθηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και δεν διέπονται επομένως πριν τη θέση σε ισχύ της οδηγίας και επομένως δεν μπορούν να διέπονται από αυτήν την νομολογία. Εμείς ζητούμε μία σειρά από μέτρα τα οποία θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει να ε, ζητήσει. Ο Πιερ Πάολο Βόλπε έχει εξηγήσει άλλωστε και τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει. Ε, και ε, επίσης ε, να αναφέρω ότι στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας 47 καθώς 31 ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επομένως δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο και στην προκείμενη περίπτωση. Ευχαριστώ. Signora Presidente, Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έδινε, δίνει τη δυνατότητα στην κυρία Κοργκόλ και στον κύριο Λουντοβίκο ε, να παρουσιάσουν τις ε, ε, περιπτώσεις τους. Εγώ δεν μιλάω σαν ε, δικηγόρος ε, της Ματζένα Κοργκόλ και του Πασκουαλίνου Λουδοβίκο. Μιλάω σαν ε, ε, Ιταλός πολίτης, γιατί εγώ ως δικηγόρος πρέπει να πω ότι έχω αποτύχει, κυρία Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές. Μαζί με τον συνάδελφο Σέρτζο Γκαλεάνο συμμετείχαμε μαζί και με άλλους Ιταλούς δικηγόρους Ε, συμμετείχαμε στην λεγόμενη απόφαση Μάσκολο της 26ης Νοεμβρίου του 2014. Εκεί αναφέρθηκαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προκείμενη περίπτωση ε, βοήθησε τους εργαζόμενους τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση και μη. Ε, εκεί το δικαστήριο αποφάσισε ότι και στην περίπτωση της εκπαίδευσης αλλά και εκτός αυτού του πεδίου, δηλαδή οι εργαζόμενοι στην υγεία, οι εργαζόμενοι στην έρευνα, στα ε, πανεπιστήμια κτλ. Ε, είπε ότι πολύ καλά έκανε το δικαστήριο της Νάπολης ε, όταν αποφάσισε ότι η σύμβαση θα έπρεπε να τροποποιηθεί και να γίνει αορίστου χρόνου. Η εφαρμογή αυτής της απόφασης σήμαινε ότι ε, σέβεται ε, την αρχή της θεμητής και καλής συνεργασίας η Ιταλική κυβέρνηση, διότι διότι ε, αυτό το θέμα είχε παρουσιαστεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ε, η βουλευτής κυρία Ρίτα Μπορσελίνο ρώτησε πώς είναι δυνατόν το 2010 ήδη ε, οι συμβασιούχοι της εκπαίδευσης δεν είχαν μονιμοποιηθεί. Και η Κομισιόν τότε είπε ότι αυτό δεν ισχύει γιατί η Ιταλική κυβέρνηση είχε διασφαλίσει ότι ούτως ή άλλως πράγματι και βάσει της απόφασης και βάσει της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έπρεπε οπωσδήποτε να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Όταν η Κομισιόν κατάλαβε ότι αυτό δεν είχε συμβεί, ξεκίνησε μια διαδικασία επί παραβάση η διαδικασία επί παραβάση ε, ξεκίνησε ε, με ε, μία επιστολή προς τον συνάδελφο Γκαλεάνο ήδη τον Αύγουστο του 2013 και εκεί ανέφερε η Κομισιόν ότι πλέον αυτή η δέσμευση θα, και η υποχρέωση δεν θα αφορούσε μονάχα τον εκπαιδευτικό τομέα αλλά και όλα, όλους τους υπολείπους και επομένως ε, και το, ε, ε, το τεχνικό προσωπικό κτλ. Όμως πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για, οποιασδήποτε, για οποιαδήποτε παιδεία εκτός το, των σχολείων δεν τροποποιήθηκαν οι συμβάσεις και στην υπόθεση Παπαλία και στις υποθέσεις Μάσκολο ε, ε, και ε, ευρεία δεν κατεγράφησαν οι καταχρήσεις αλλά δεν, δεν εφαρμόστηκε ε, η αρχή της αυτόματης μετατροπής της σύμβασης από ορισμένου χρόνου ε, σε αορίστου μετά τους 36 μήνες. Τι έγινε από εκεί και πέρα και ένα όλες αυτές οι αποφάσεις ήταν υπέρ των εργαζομένων. Τι έγινε δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω. Ε, εν προέκυψε ε, η νομοθεσία για την απασχόληση των νέων ε, η οποία φέρει το όνομα Jobs Act και εκεί ανακαλύψαμε ότι ε, η Jobs Act εξαφάνιζε κατά κάποιο τρόπο την αντίστοιχη οδηγία του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην απόφαση 362 του 2013, γνωστή ως, ως ε, υπόθεση Φιαμίνγκο του Ιουλίου 2014, η Κομισιόν ε, ζητήθηκε να παρέμβει. Σε αυτή την περίπτωση όμως η Κομισιόν δεν έκανε παρέμβαση εναντίον της ε, κυβέρνησης της Ιταλίας, δηλαδή δεν έκανε παρέμβαση με διαδικασία επί παραβάση κατά της της Ιταλικής κυβερνήσεως αλλά ξεκίνησε με διαδικασία επιπαραβάση εναντίον του Λουξεμβούργου. Δεν είναι δυνατόν όμως να ε, ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν ξαφνικά να εξαφανιστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία από την Ιταλική Ένωμη Τάξη. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν είναι δυνατόν. Ε, εμείς έχουμε την απόφαση Κομισιόν κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ε, του 2015 και δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι ε, μονάχα το Λουξεμβούργο δεν έχει σεβαστεί την οδηγία 9970 και δεν ξέρουμε καν αν υπάρχουν και πόσοι είναι αυτοί οι συμβασιούχοι από το Λουξεμβούργο. Δεν καταλαβαίνουμε ε, γιατί η Κομισιόν αρχιοθέτησε τη διαδικασία 21-24. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση μάσκολο, από τη στιγμή που είναι υποχρεωτική η τροποποίηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, δεν είναι δυνατόν λέω να συμβαίνει αυτό και ο κύριος Λουντοβίκο να υποχρεώνεται να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δεν μπορεί να βρει το, χρόνο, το, το δίκιο του. Κοιτάξτε, εγώ ζητώ να παρεύει το Κοινοβούλιο μέσω ψηφίσματο. Πάω λίγο παραπέρα από ότι οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Να κάνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό, γιατί αφορά και την Ισπανία και αφορά και άλλε χώρε. Δεν αφορά μονάχα την Ιταλία. Η οδηγία είναι οδηγία και είναι και κοινωνική συνθήκη. Δεν είναι δυνατόν μετά από 50 αποφάσεις του δικαστηρίου που έχουν ερμηνεύσει την οδηγία 90-70 ε, ε ξανά αναρωτιόμαστε και ξύνουμε το κεφάλι μας για να δούμε αν θα εφαρμοστεί αυτή η 90-70 και αν υπάρχει παράβαση ενώ ξέρουμε ότι έχει παραβιαστεί αυτή η οδηγία από την Ιταλική κυβέρνηση. Εμείς ως πολίτες Ευρωπαίοι, ως πολίτες της ε, Ιταλίας έχοντας συνεργαστεί ε, με ευρωπαϊκές αρχές ε, όταν φτάσαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζήτησαμε ζητούμε από την Επιτροπή σας, εδώ την Επιτροπή Αναφορών, ε, να ε, ε, μας υποστηρίξει για την, για την για ε, να ξεκινήσει διαδικασία επί παραλήψη ε, για την αρχιοθέτηση της ε, υπόθεσης αυτής. Γιατί εάν είχε συνεχιστεί η υπόθεση και αν η Κομισιόν δεν είχε αποσυρθεί, τότε δεν θα είχαν προκύψει όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. One Μπορώ να απαντήσω αμέσως σε ένα σημείο. Σήμερα το πρωί αποφασίσαμε να έχουμε δημόσια ακρόαση για ακριβώς αυτό το θέμα. Το φθινόπωρο εδώ στην Επιτροπή μας. Είναι λοιπόν απολύτως κατάλληλη στιγμή και με χαρά σας το ανακοινώνω αυτό. Δεν θα χρειαστεί να έρθετε στις Βρυξέλλες. Ε, μπορείτε από την Ιταλία, από τον υπολογιστή σας να παρακολουθούσετε την ακρόαση αυτή, διότι θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο η ακρόαση, όπως άλλωστε και η σημερινή συνεδρίαση. Όλοι σας λοιπόν, οι συναδελφοί σας και ελπίζουμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και άλλοι εμπειρογνώμονες πανεπιστημιακοί σε όλη την Ευρώπη να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο από όπου και να βρίσκονται την ακρόαση αυτή. Με χαρά σας το ανακοινώνω αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά και η μόνη ακρόαση που θα κάνουμε το απόγευμα, ε, το φθινόπωρο θα έχει ακριβώς αυτό το θέμα να απευθυνθώ τώρα στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ιταλίας και τον εκπρόσωπό της, τον κύριο Μαουρίσιο Ανδράκιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ αρχής να πω ότι η παρέμβασή μου θα, έχει, θα είναι γενικού χαρακτήρα. Γιατί όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε πέντε προδικαστικά ερωτήματα κατά της ε, ε Ιταλίας ε, που λένε περίπου το ίδιο πράγμα. Δηλαδή την ε, καταχρηστική ε, ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ε, διακριτική μεταχείριση εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου και αορίστου κτλ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ε, υπογραμμίσω τον τρόπο με τον οποίο ε, η Ιταλική ε, κυβέρνηση προτίθεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και σε συμφωνία βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λύσει αυτά τα επίδικα αντικείμενα. Πρώτον, τροποποιώντας την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα δημόσιας διοίκησης, δηλαδή απασχόλησης στο δημόσιο και επίσης να πάρει και προληπτικά μέτρα μέτρα έτσι ώστε ε, να λυθούν, να σταματήσουν αυτές ε, οι καταχρήσεις που ε, σχετίζονται με τη συμβάση ορισμένου χρόνου και επίσης την πρόθεση της Ιταλικής κυβέρνησης λέω να λάβει κυρώσεις έναντι των αρχών οι οποίες έχουν αυτήν την πρακτική των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Όσον αφορά τώρα την ε, διακριτική μεταχείριση που ανέφεραν οι εργαζόμενοι, διάκριση μεταξύ εργαζόμενων με σύμβαση ορισμένου και ορίστου χρόνου, ε, έχει αποφασιστεί ε, ότι θα ξεκινήσει η συλλογική διαπραγμάτευση ε, και διαβούλευση ε, με τους εργαζόμενους έτσι ώστε να οριστεί πλέον και δια νόμου η μη διακριτική μεταχείριση εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου και αορίστου χρόνου. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να εξηγιανθεί κατά κάποιο τρόπο αυτός ο βόρβορος. Ευχαριστώ πολύ. Let's all hope that this will happen soon. Ελπίζουμε όλοι να συμβεί αυτό και μάλιστα όσο γίνεται πιο σύντομα. Ήδη έχει καθυστερήσει πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τένα Θερμαζάμενα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τις καταστάσεις που περιγράφουν οι αναφέροντες στην Ιταλία και έχει στείλει ε, αιτήματα για περισσότερες πληροφορίες στις Ιταλικές αρχές. Ε, εξετάζουμε ακόμα την υπόθεση. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις ε, σχετίζονται με τις διακρίσεις που γίνονται στον δημόσιο τομέα της Ιταλίας και όλοι μας περιμένουμε μια πολύ σημαντική απόφαση στο θέμα αυτό διότι έχει παραπευθεί η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2016 από Ιταλικό Δικαστήριο. Το Δικαστήριο ζητάει κατευθυντήριες γραμμές ε, όσον αφορά την αποζημίωση σε περίπτωση κατάχρησης ε, λόγω διαδοχικών ε, συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Μόλις λάβουμε την απόφαση αυτή θα αποφασίσουμε σχετικά με τα επόμενα μας βήματα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, πολύ σύντομη απάντησή σας. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κυρία Κούνεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάχρηση των προσωπικών συμβάσεων εργασία από φορεί στο, δημόσιο τομέα δεν μα ξαφνιάζει. Το γνωρίσαμε και εμεί στην Ελλάδα πολύ καλά έγιναν πολλοί αγώνε των εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου χρόνου που αν και ικανοποιούσαν βάγιες και διαρκείς ανάγκε, δούλευαν με συμβάσει ορισμένου χρόνου τρία, τέσσερα, ακόμα και δεκαπέντε χρόνια με μικρές διακοπές. Το κράτος και το δημόσιο επιχρόνια λειτουργούν σαν τους χειρότερους εργοδότες. Μας ξαφνιάζει η καθυστέρηση της Επιτροπής Πώς είναι δυνατό να εκκρεμεί τόσα χρόνια η εφαρμογή της αποφάσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και η Κομισιόν να μην κάνει τίποτε και να ελέγξει, για να ελέγξει εάν ενσωματώνεται μια οδηγία στην εθνική νομοθεσία. Η Κομισιόν πιθανότατα ελέγχει επιμελώς την ενσωμάτωση των οδηγιών στην εθνική νομοθεσία, διότι όπως φαίνεται από τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων, οι εθνικοί νόμοι αφήνουν παρατηράκια που επιτρέπουν σε δημόσιες αρχές να παρακάμπτουν την οδηγία στην ουσία της. Ένα δικό μας παράδειγμα στην Ελλάδα είναι οι αναπληρωτές κατοικητές που τοπικά είναι μη συνεχίσει οι του με αποτέλεσμα για χρόνια οι κατοικητέ να καλύπτουν με τρίμηνα διαλύματα. Άλλο τρόπο καταστρατηγική είναι οι συμβάσεις έργο, π.χ. οι καταρρίστρες Υπουργείου Οικονομικών, επί 19 χρόνια. Εδώ το θέμα που εξετάζουμε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών δεν αφορά μόνο μια περίπτωση όπως φαίνεται. Έχουμε πάνω από 20 αναφορές μόνο από Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία που αφορούν χιλιάδες οικογένειες. Να φανταστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι συμβαίνει. Πόσο είναι δεδομένο αυτό το φαινόμενο σκλήρης εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Η εργασιακή ανασφάλεια, η επισφαλής της εργασίας συνδέονται σε πολλές χώρες με την κατάχρηση που κάνουν οι κυβερνήσεις στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που στην πραγματικότητα μετατρέπεται σε πολιτικό παζάρι και σε ομοιρία. Για αυτούς τους λόγους προτείνω να μείνει ανοιχτή αναφορά νούμερο 13, να σταλεί επιστολή προς την Ιταλική κυβέρνηση η οποία να εξηγεί τους λόγους που συνεχίζει την καταχρηστική χρησιμοποίηση των διαδοχικών συμβάσεων, να προχωρήσουμε στην ανατέτηση μελέτης και ενδεχομένω και ακροάσει στην Επιτροπή Αναφορών για την κατάχρηση των συμβάσεων εργασία ορισμένων χρόνων, όπω μα είπατε ότι έχει γίνει η οργάνωση πια. Αλλά οπωσδήποτε να προχωρήσουμε ως Επιτροπή στην κατάθεση προφορικής ερωτήσης και ψήφισμα προς την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όπως μας πρότειναν και οι καταγγέλνοντες. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο στον κύριο Μπέκερ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί, έχουν ήδη εκφραστεί. Είναι σαφέστατο το ότι χρειάζεται δράση Και εξ όσων γνωρίζω και εξ όσων έχω διαβάσει στις εκθέσεις της Γραμματείας για τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρώ ότι η Επιτροπή έχει δράσει, δρά και είναι ευθυγραμμισμένη. Δεν βλέπω κανένα έλλειμμα στη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να είμαι ειλικρινής. Από ό,τι μαθαίνω όμως από τις λεπτομέρειες, για παράδειγμα για την αναφορά 4, 11, 13, 22, 4, 29, για αυτές τις αναφορές ακόμα ε, και οι αποφάσεις του δικαστηρίου εκκρεμούν, Άρα θα πρέπει να περιμένουμε ε, ενημέρωση για τη σχετική πρόοδο, ενώ για τις αναφορές 988 και 216, 1026 και 1063, το συγγνώμη, 1026 και 1063 του 2016 δεν έχουμε καθόλου λεπτομερή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το περιμένουμε και αυτό. Και τις προωθούμε τις αναφορές ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σχολιάσει και εκείνη για ένα θέμα που την αφορά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σαφές ότι όλες αυτές οι αναφορές πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, η πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Ελεονόρα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αναφέροντες που βρίσκονται σήμερα εδώ, έτσι ώστε να καταγγείλουν αυτήν την κατάσταση. Συγκλονίστηκα από την συντομία της απάντησης της Κομισιόν, αλλά και από αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της ε, μόνιμης αντιπροσωπείας της Ιταλίας, ε, ο οποίος με ένα «ελπίζουμε ότι θα» ε, με μία μονοκοντιλιά λοιπόν έσβησε το θέμα. Δεν είναι δυνατόν να βασιστούμε σε ε, ε, υποσχέσεις και γι' αυτό λοιπόν καταγγέλουμε την κατάσταση και ε, συμφωνούμε ότι οι, οι αναφέροντες καταγγέλουν καταστάσεις οι οποίες διαρκούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταχρήσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν σταματήσει ε, και βεβαίως αυτό είναι ευθύνη πολλών κυβερνήσεων διαδοχικών της Ιταλίας αλλά και ευθύνη οπωσδήποτε και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με πολύ επιφανειακό τρόπο έκανε τη δουλειά της και αναφέρομαι και στην, ε, ε, στην 21-24 του 2010. Αν είχε γίνει για το Δημόσιο Σχολείο, αν είχε γίνει ε, καλά και σωστά η δουλειά της Κομισιόν, τότε η Κομισιόν θα είχε ήδη καταλάβει ότι ε, στο, στην εκπαίδευση είναι εκατοντάδες οι καταχρήσεις ε, και χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, βρεθεί με επισφαλείς θέσεις εργασίας. Κατά την άποψή μου λοιπόν εδώ έχουμε απέναντί μας ανθρώπους οι οποίοι καταγγέλουν τον εφιάλτη της επισφαλούς ε, εργασίας, τον εφιάλτη του να ζουν ε, χωρίς ε, να ξέρουν ποιο είναι το μέλλον τους. Αφορά το θέμα αυτό πάρα πολύ την Ιταλία και γι' αυτό πραγματικά η παρέμβασή μας να είναι η παρέμβαση από πλευράς των αρχών και των Ιταλικών και των Ευρωπαϊκών. Η παρέμβαση αυτή λέω να είναι ισχυρή έτσι ώστε να σταματήσει και η διάκριση μεταξύ ε, των ε, εργαζομένων στο δημόσιο τομέα με συμβάσεις εργασίας ε, ορισμένου και ορίστου χρόνου. μπορεί να έγιναν, μάλλον θα πρέπει να γίνουν και όλοι, όλες οι νομοελεγκτικές διαδικασίες έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα γίνουν καλά. Νομίζω ότι είναι σαφές ε, ότι και από πλευρά της Κομισιόν και από πλευρά της ιταλική κυβέρνησης ήταν ελιπέσταση, ελιπέστατη η πρόθεση εξέβρεσης λύσης και επομένως ε, πραγματικά χαίρομαι ε, που όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν ότι πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό. Θα πρέπει να ρίξουμε τους προβολείς του Κοινοβουλίου κατά κάποιο τρόπο στο θέμα αυτό. γιατί ε, πραγματικά το λέω και το επαναλαμβάνω, εδώ παίζεται το κεφάλι και η ζωή εκατοντάδων ε, χιλιάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους, ε, από την, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από την Πορτογαλία. Ακούσαμε πριν από λίγο την περίπτωση της Ελλάδος. Επομένως, νομίζω ότι είναι σαφές ότι ζητούμε να μείνουν ανοιχτές όλες αυτές οι αναφορές και να δώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα απαντήσεις τους αναφέροντες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοράου, ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι μέλος αυτής της επιτροπής ε αλλά ξέροντας ε, ότι θα ε, γινόταν λόγος ε, για αυτές τις επισφαλείς θέσεις εργασίας και μια και είμαι και εκλέγομαι άλλωστε και στην Σικελία, πραγματικά έπρεπε να έρθω να ακούσω τι έχουν να πούν οι αναφέροντες και δεν μπορούσα να μην πάρω και το λόγο, γιατί είναι σαφές ότι εδώ μιλάμε για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, κυρία Πρόεδρε, το ξέρετε ότι επανειλημμένα έχουμε μιλήσει για θεμελιώδη δικαιώματα, για δικαιώματα ανθρώπων που ζουν μάλιστα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία η οποία δεν έχει ε, εφαρμοστεί από μία από τις πιο μεγάλες ας πούμε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, απ' την άλλη πλευρά η Κομισιόν η οποία ξέρει πολύ καλά να κουνάει το δάχτυλο όταν κάτι δεν πάει καλά ας πούμε στους προπολογισμού ε, ή και στον προπολογισμό τη Ιταλία, εδώ με μία μονοκοντιλιά και με μία ε, λέξη το ξεπέταξε το θέμα. Εντάξει, καταλαβαίνω και τον εκπρόσωπο της ε, Ιταλική μόνιμη αντιπροσωπεία. καταλαβαίνω την αμηχανία σα πρόκειται για μια κατάσταση η οποία έχει εγκατασταθεί εδώ και 10-15 χρόνια. Ε, και είναι λίγο δύσκολο. Εδώ ε, μιλήσαμε προηγουμένως ε, για 18η, 19η ανανέωση ε, συμβάσεις ορισμένου ε, χρόνου. Αλλά ξέρετε εδώ δεν μιλάμε για ανανέωση ε, ας πούμε της κάρτας οπαδού μιας ομάδας ή της μιας οποιασδήποτε διαδικασίας έτσι, συμμετοχή σε ένα, μια λέσχη σε κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε για χρόνια πολλά. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν ξέρουν πώς θα στείλουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο, αν θα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο. Τι να σας πω, δεν ξέρω εάν ε, ε, μπορεί να μας πει η συνάδελφος Όγκαν ε, εάν κάτι παρόμοιο γίνεται στη Δανία ή ο κύριος Μπέκερ να μας πει αν γίνεται κάτι αντίστοιχο στην Αυστρία. Και εν πάση περιπτώσει εγώ στρέφομαι προς την Κομισιόν και λέω εδώ μιλάμε για κάτι ειδικό το οποίο έχει μεγάλο πολιτικό βάρος στην ουσία. Αυτοί οι άνθρωποι με το σύστημα αυτό έχουν κρατηθεί όμοιροι από μία ε, ε, ε, πολιτική τάξη στην Ιταλία η οποία χρησιμοποίησε αυτό το σύστημα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και των συμβασιούχων και το γεγονός ότι δεν προβλέπονται ε, μηχανισμοί νομοθετικοί που να αποτρέπουν τη δημόσια διοίκηση να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους ε, εργαλεία. Γιατί εδώ δεν μιλάμε ε, για μεμονωμένες επιλογές, μιλάμε για κεντρικές πολιτικές επιλογές. Εκεί λοιπόν πρέπει ο πολίτης να δει ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι δυνατή η τελική κυβέρνηση και η, συγγνώμη, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ακριβώς τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει ότι πρέπει να σταματήσει η κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και ευχαριστώ και την συνάδελφο Εύη, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και εσά, κυρία Πρόεδρε ε, που αναφερθήκατε στην ακρόαση. Ναι, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να ακουστεί το θέμα αυτό, να συζητηθεί και στην Ολομέλεια. Αφορά πάρα πολλού πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες χώρες. και δεν θα τις απαριθμίσω, θα έχουμε άλλωστε την ακρόαση. Είναι όμως δραματικό θέμα και στην Γερμανία υπάρχουν αντίστοιχε καταχρήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση για την ακρόαση που θα έχουμε. Πρόεδρος, έτσι κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών μας και ε, ξαναδίνω το λόγο στους αναφέροντες δύο λεπτά ο καθένας. Έχουμε χρόνο. Εάν θέλετε. Εάν δεν θέλετε, θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Πιέρ Παύλο Βόλπε, παρακαλώ. Allora, la Είναι, μας προκαλεί αμηχανία αυτή η απάντηση της Ιταλικής κυβέρνησης, του εκπροσώπου δηλαδή. Για μία ακόμα φορά χρησιμοποιεί την ε, κύρωση ε, ε, σαν αποτρεπτικό μέσο, ενώ ούτε η Ρήτρα ούτε η οδηγία προβλέπει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει η τελική κυβέρνηση ε, να ορίσει κάποια μέτρα τα οποία θα είναι ενεργητικά, τα οποία θα είναι σαφή, τα οποία θα είναι ακριβώς περιγεγραμμένα, έτσι ακριβώς όπως ορίζουν οι αποφάσεις των δικαστηριών. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η κύρωση προς τους υπευθύνους είναι αποτρεπτική. Ε, το είπε άλλωστε και το ίδιο το δικαστήριο. Και εμείς αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ένα και έχουμε στείλει εκατοντάδες ε, καταγγελίες και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και δεν μπορώ να το βάλω στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η Κομισιόν μία διαδικασία ε, επιπαραβάση σχετικά με με διακριτική μεταχείριση. Τι κάνουμε εδώ πέρα, περιμένουμε τον κοντό, δεν κατάλαβα. Τι συμβαίνει εδώ. Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα μία διαδικασία επιπαραβάσει. Από τον Νοέμβριο του 2014 ε, εκδόθηκε η απόφαση Μάσκολο και αμέσως θα έπρεπε η Κομισιόν να ξεκινήσει ε, και να καταθέσει έναντι της Ιταλίας διαδικασία επί, παραβάση, ε, συγγνώμη, επί παραλήψη. Και ακόμα την περιμένουμε. Και ποια είναι αυτή τώρα η μεταρρύθμιση που θα ξεκινήσει δίθεν η Ιταλική κυβέρνηση έτσι ώστε να εξηγηθεί η κατάσταση και έτσι ώστε να μην υπάρξει διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ε, τους εργαζόμενους που έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και αυτούς που έχουν ε, ορίστου. Τίποτα, μηδέν. Καμία μεταρρύθμιση, αυτό έχω να σας πω. Καμία απολύτως. Και έπειτα θα πρέπει να δούμε την ρήτρα 5, δηλαδή τις αντικαταχρηστικές και προ... τα αντικαταχρηστικά προληπτικά μέτρα. Ε, ακόμα και στη μεταρρύθμιση Μπαντία δεν προβλέπεται καμία ε, τροποποίηση. Υπάρχει μάλιστα δε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που λέει ότι για μία ακόμα φορά, ακόμα και με την ε, και με τη μεταρρύθμιση Μπαντία και λαμβάνοντα υπόψη όλες τις αποφάσεις του δικαστηρίου, τίποτα δεν κάνει η Ιταλική κυβέρνηση. Τι κάθεται, κάθεται και ξύνει το κεφάλι της, λέει ο μιλήτης, έτσι ώστε να μπορέσει να βρει κάποια λύση. Δήθεν, δήθεν. Ε, Δηλαδή αυτό το άρθρο 97 που είναι το τοτέμ και το προσκυνάμε όλοι του συντάγματος να το σκίσουμε, να το κόψουμε, να τα κάνουμε κομματάκια γιατί δεν μας δεν, δεν, δεν, το χρησιμοποιεί κανένας. Και έχουμε και την απόφαση Τσάρα του 15. Ε, αυτό πρέπει να κάνει η, η Ιταλική κυβέρνηση. Ένα πράγμα πρέπει να κάνει. Πρέπει να σταματήσει αυτήν την επισφάλεια. Πρέπει να σταματήσει αυτές τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ελίσαντε Ματέο, παρακαλώ. Io volevo soltanto fare delle precisazioni, soprattutto con dei riferimenti non... Εγώ θα ήθελα να αναφέρθω σε αυτά που είπε ο εκπρόσωπο της τελικής κυβέρνησης. Αναφέρθηκε στο νόμο του 2001 την 448. Εκεί, ε, σε αυτήν θέλω να κάνω εγώ αναφορά, εκεί αναφέρεται ακριβώς ότι η περιφέρεια της Σικελίας και οι φορείς του ε, θα πρέπει να μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου βάση του, ε, του νόμου 61. Επίσης ανεφέρετο ότι ε, οπωσδήποτε θα έπρεπε τα χρήματα αυτά ε, τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να αντιληθούν από το άρθρο 61 της χρηματοδότησης υπεριθμών 1 31 31 1941 για την περιφέρεια της ΕΣΥ και Ελίας. Η ομιλήτρια δυστυχώς πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, είναι αδύνατο να καταγραφούν όλοι οι αριθμοί. Ε, στο άρθρο 1 λοιπόν αναφέρεται σαφώς ότι ε, για να μην σταματήσουν ε, οι θέσεις οι οποίες καλύπτονται κυρίως όσον αφορά ε, την αποχέτευση, την δημόσια υγεία, τις, τις θέσεις εργασίας για την δημόσια διοίκηση θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι οι εργαζόμενοι να, καλύπ, να, έχουν θέσεις και συμβάσεις ε, ο αορίστου χρόνου. Ε, ακόμα όμως τώρα περιμένουμε μια σταθεροποίηση της ε, κατάστασης. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2016 ο κύριος Μπαρναμπά, ο δικός μου δηλαδή, ε, ο, ο αναφέρον τον οποίον εγώ ε, εκπροσωπώ, ε, για μία ακόμα φορά πήγε στην περιφέρεια της Σικελίας όπου πάλι δεν βρήκε το δίκιο του, γι' αυτό δεν έχουμε καμία απολύτως διάθεση να πιστέψουμε αυτά που μας λέει η τελική κυβέρνηση. Η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν ε, ε, υπήρξε καμία προστασία ούτε από, τη δικαστή, από τις δικαστικές αρχές, ούτε από πουθενά αλλού. Ε, ε, όπως σας είπα προηγουμένως, ε, η πρώτη ακρόαση ορίστηκε για τον πελάτη μου δύο χρόνια μετά από την κατάθεση της, του, της υπόθεσής του. Στην ουσία όμως και οι δικαστές στην Κατάνια αποφάσισαν ότι η αποζημίωση θα ήταν αντίστοιχη με το εισόδημα 8 μηνών. Μα τι να κάνουν 8 μήνες μπροστά στη ζημία που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι. Επομένως, όταν από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ε, ότι ε, ναι, έχουμε ακόμα μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και αυτό δεν αρκούσε. Και όταν από την άλλη μεριά έχουμε και τον εκπρόσωπο της Ιταλικής κυβέρνησης να λέει ναι, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει. Και από την τρίτη πλευρά έχουμε το δικαστήριο το οποίο ορίζει πρώτη ακρόαση ε, δύο και τρία χρόνια μετά. Καταλαβαίνετε ότι θα έχει ολοκληρωθεί η, ο εργασιακός βίος αυτών των συμβασιούχων και θα είναι έτοιμοι να πάρουν τη σύνταξή τους. Ε, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει η κατάσταση αυτή. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, οι συμβασιούχοι, κάποια στιγμή να καλύψουν τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαρία Κάρμελα Τιματέα. Κυρία Πρόεδρε, ε, οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν πολύ σωστά στο θέμα αυτό. Ε, Λοιπόν, λέγαμε ότι η πρώτη ακρόαση, η πρώτη μελέτη τέλο πάντων του θέματο ενώπιον του δικαστηρίου έχει οριστεί για δύο χρόνια μετά την κατάθεση ε, των εγγράφων. Αλλά για να έχουμε την πρώτη απόφαση θα περάσουν έξι και 7 και 8 χρόνια. Επομένω, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο είπαν προηγουμένως λίγο και οι συνάδελφοι. Ήδη εδώ η απόφαση που δόθηκε ε, από την Ιταλική κυβέρνηση είναι απαράδεκτη ε, και ε, παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πουθενά δεν λέει ότι θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις οι οποίες να είναι αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση, προβλέπεται πουθενά ε, να υπάρξουν προληπτικές και αποτρεπτικές ε, κυρώσεις. Ε, ε κοιτάξτε, εγώ ξέρω, μια, εγώ ξέρω ότι γνωρίζω από παιδάκι την, την πελάτηδα, πελάτησά μου και τώρα είμαι ο δικηγόρος της και αυτή από όσα χρόνια τη γνωρίζω ήταν στην ίδια θέση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ευχαριστώ. Ο κύριο Σέρτζο Γκαλιάνο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίω εγώ συμφωνώ απολύτω με όσα είπαν ε, οι στην συναδελφοί μου σχετικά με την ανεπάρκεια της απάντησης και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πλευρά του εκπροσώπου της τελική κυβερνήσεω. Ε, θα ήθελα για να, για να ολοκληρώσουμε λίγο την εικόνα να σα πω ότι το 2016 ο Άριος Πάγος ε, πήρε μια σειρά αποφάσεων. Δηλαδή, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία η παραβάση από πλευρά τη Κομισιόν ε, και έθεσε δύο ερωτήματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, α, ποιος ε, ε, ε, ε, ποιος μπορεί να δώσει τελειωτική λύση. Μάλλον ότι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους, έχουν σταθεροποιηθεί λέει ο μιλητής, τότε λέει ο Άριος Πάγος δεν έχουν δικαίωμα σε αποζημίωση. Δηλαδή Δηλαδή, ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει δυνατότητα αποζημίωσης, ε, ενώ ο ιδιωτικός υπάλληλος στην Ιταλία έχει δικαίωμα, ο οποίος έχει υποστεί κατάχρηση, έχει... Ε, έχει την δυνατότητα να αποζημιωθεί ε, με ποσό αντίστοιχο από 2,5 μέχρι 12 μήνες. Επομένως εδώ έχουμε διακριτική μεταχείριση. Ε, δηλαδή, ε, όταν ε, ο εργαζόμενος στο δημόσιο μονιμοποιείται, τότε ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο ή έρεται η διαφοροποίηση και η διακριτική μεταχείριση που είχε. Όμως αυτό δεν πρέπει να ισχύει με την έννοια ότι πρέπει και να σταθεροποιηθεί, δηλαδή πρέπει και να βρεθεί η σταθερή θέση απασχόλησης, αλλά και να αποζημιωθεί για την προηγούμενη κατάσταση. Τι συμβαίνει όμως, οι εργαζόμενοι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έχουν ε, επιτύχει αποζημίωση ε, ε, θα πρέπει τα προηγούμενα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει σύμφωνα με την απόφαση του Αρίου Πάγου να επιστρέψουν τα χρήματα. Αυτό όμως αντιτίθεται στην, Ευρωπαϊ... στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Μάσκολο. Κάποιος που δουλεύει στο σχολείο, ας πούμε, πρέπει ο ίδιος ε, να αποδείξει ότι καλύπτει μία καινή θέση. Ενώ ε, ενώ ε, υπάρχει ήδη η υποχρέωση του εργαζόμενου, του εργοδότη, εν προκειμένου του Υπουργείου Παιδείας, ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει καινή θέση. Ε, αυτό σημαίνει αντιστροφή της ε, ε, υποχρέωσης της απόδειξης και αυτή η κατάχρηση είναι πρόδειλη. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει κενή θέση και την καλύπτει. Επίσης, τελειώνοντας να πω ότι στη Σικελία υπάρχουν κάποιες κοινότητες οι οποίες Ε, υπάρχουν, λέω, κοινότητες ε, οι οποίες ε, κοινοποιούν, ας πούμε, στο διαδίκτυο το οργανόγραμμά τους και στους 200 υπαλλήλους βλέπεις ότι έχουν 150 συμβασιούχους και 50 μονίμους. Αλλά αυτοί οι 150 κάθε χρόνο είναι οι ίδιοι συμβασιούχοι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Επίσης, να μην λησμονούμε ότι εάν αυτοί οι συμβασιούχοι κάποια στιγμή έφευγαν, αφαιρούνταν από την δημόσια διοίκηση, τότε το δημόσιο οικοδόμημα θα κατέρεε. Ευχαριστώ. Ε, ε, Κυρία Πρόεδρε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τις σύντομες ε, είναι η αλήθεια παρεμβάσεις της εκπροσώπου της Κομισιόν και του εκπροσώπου της Ιταλικής Κυβερνήσεως. Εμείς Ελπίζαμε να έχουμε κάτι παραπάνω από την Κομισιόν, γιατί ο κύριος Γκαλεάνο και ο υποφαινόμενος εκπροσωπούν την κυρία Σαντόρο στην ε, ε, υπόθεσή της ενώπιον του δικαστηρίου του Τράπανο. Περιμέναμε δε την μετάφραση των γραπτών παρατηρήσεων, μεταξύ των οποίων και την νέα θέση της Κομισιόν. Εάν τα είχαμε τα στοιχεία αυτά, θα καταλαβαίναμε γιατί σταμάτησε η Κομισιόν τη διαδικασία επί παραβάση της Κομισιόν, ε, απλώς υποβάλλοντας για μία ακόμα φορά ένα προδικαστικό ερώτημα. Δεν είχαμε όμως κάτι τέτοιο, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να ευχαριστήσω την Κομισιόν, ε, την Επιτροπή σας μάλλον, ε, για, την, ε, για τη συζήτηση. Και να σας πω το εξής. Ο κύριος Φέρνοντ, δικαστής Σουηδός, δικαστή στην υπόθεση Βαλέντσα και λοιπόν της 18ης Δεκάτου 2012. Ο δικαστής μαζί με το κολέγιο του δικαστηρίου που είναι ίδιο με το κολέγιο της απόφασης Μάσκολο απεφάνθη ότι πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης ακόμα ε, και ε, σε αυτούς και για αυτούς που μέσω συστάσεων ε, έγιναν, υπέγραψαν συμβάσεις και προσελήφθησαν και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί σωστά το, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, δηλαδή στους Σικελούς, στο σχολείο, στην ε, διοίκηση, ε, σε όλους αυτούς που ε, προσελήφθησαν μέσω ασέπα, το πούμε, μέσω ε, εξετάσεων. Ε, ε, αυτοί οι άνθρωποι δεν πήραν ποτέ συμβόλαια, συμβάσεις αορίστου χρόνου. Και τότε ο δικαστής, ο Σουηδός, είπε εντάξει, μα σταματήστε πια να λέτε και να ξαναλέτε τα ίδια πράγματα. Μα κυρία Πρόεδρε, στην περίπτωση Παπανία είχαμε 30 χρόνια 30 χρόνια ε, τον άνθρωπο αυτό, τον κύριο Παπανία, ο οποίος ε, ε, ήταν για 30 χρόνια συμβασιούχος δάσκαλος μουσικής. Τώρα τι να σας πω εγώ. Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, έχει για 30 χρόνια οργανώσει ε, την ε, φιλαρμονική της πόλης του, της ΑΟΣΤΑ, προφανώς κάποιο δικαίωμα θα έχει έτσι ώστε να μονιμοποιηθεί. Τώρα, μας έχει υποθεί επανειλημμένα ε, ότι η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, τα κράτη γενικά της Ευρωελάδα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μονιμοποιήσουν πρέπει να έχουν χρήματα, πρέπει να επενδύσουν. Και ό,τι δήθεν λόγω έλλειψης πόρων δεν, δεν υπάρχει μονιμοποίηση. Αλλά στις 26 Μαρτίου του 2014, στην υπόθεση Μάσκολο, εμείς δώσαμε τα δικά μας εσωτερικά ε, στοιχεία της εφορίας και του ελεγκτικού συνεδρίου, βάσει των οποίων η μονιμοποίηση των ε, συμβασιούχων του σχολείου θα ε, είχε αποτέλεσμα ε, να αποταμιευθούν 600 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για τους συμβασιούχους του σχολείου. Τη εκπαίδευση εν πάση περιπτώσει. Τόσα θα, θα κερδίζαμε. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτό το θέμα της λιτότητας, που είναι η καραμέλα που ακούμε συνέχεια, δεν έχει καμία σχέση με τη μονιμοποίηση των... Ε, συμβασιούχων, γιατί η μονιμοποίηση των συμβασιούχων τελικά μας οδηγεί σε εξοικονόμηση όπως άλλωστε και το, η πρωτοβουλία του κυρίου Ρέντσι για την Jobs Act, όπως και η κίνηση της Κομισιόν ε, να αρχιοθετήσει την 21-22 που σας ε, ε, από της Κομισιόν ε, που, σημα, που σήμαινε στην ουσία ότι όλα πηγαίνανε καλά και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ε, και όλα καλά ε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην ουσία κάποιος λέει ψέματα. Και σας το λέω εγώ. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχοι στο σχολείο που λόγω της ελλειπούς εφαρμογής της απόφασης Μάσκολο είναι ακόμα συμβασιούχοι. Υπάρχουν ε, εκατοντάδες δε ε, ε, άνθρωποι οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν χωρίς να έχουν περάσει από κανένα διαγωνισμό, χωρίς να έχουν που, να δεν είχαν ποτέ εργαστεί στη ζωή τους και που κοστίζουν τρία δις παραπάνω στο Ιταλικό Δημόσιο. Δηλαδή στην ουσία μονιμοποιήσαμε ανθρώπους που τους πήραμε από τα σπίτια τους που καθόντουσαν ωραία και καλά και διώξαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν συμβασιούχοι για χρόνια. Επομένως δεν είναι δυνατόν ε, εμείς να ε, συμφωνήσουμε ότι για λόγους οικονομικούς ε, δεν μονιμοποιούνται οι συμβασιούχοι. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι. Ευχαριστώ. Να. Ωραία, ας προσπαθήσουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους σας που μας δώσατε τόσες πληροφορίες. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα αφήσουμε ανοιχτές όλες αυτές τις αναφορές φυσικά και περιμένουμε να λάβουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα σχετικά με τις διαδικασίες επιπαραβάση και την κατάσταση όσον αφορά κάθε μία από αυτές, γραπτός. Διότι, λυπάμαι που το λέω, αλλά η σημερινή σας απάντηση δεν αρκεί. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο εκτενής. Θα μπορούσατε να μας είχατε δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι τον Ιανουάριο του 2017, πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η Γενική Διεύθυνση απασχόληση ενημέρωσε τον αναφέροντα ότι κατόπιν αιτήματο για περαιτέρω πληροφορίες από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το θέμα αυτό, θα ε, υποβάλουν στον αναφέροντα αναλυτική απάντηση. Εμένα με εκπλήσει το ότι αυτό ούτε καν το αναφέρατε. Θα ήθελα λοιπόν αναλυτικές πληροφορίες προς την Επιτροπή μας ακριβώς σχετικά με αυτό το θέμα. Διότι δεν είμαστε εχθροί του Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Διαμεσολαβήτριας, ε, συνεργαζόμαστε και θα πρέπει να λαμβάνουμε ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες με αυτόν και να επαναλάβω ότι θα ξανασχοληθούμε με το ε, θέμα αυτό, όχι με τις αναφορές, αλλά με το θέμα ε, κατά την ακρόασή μας το φθινόπωρο και περιμένω να ακούσω και τη δική σας συνεισφορά. Κατόπιν θα δούμε τι μέτρα θα λάβουμε. Προς τις Ιταλικές αρχές και προς τους εκπροσώπους ε, της ε, μόνιμης αντιπροσωπείας, θα ήθελα να εκφράσω πολύ σοβαρή ανησυχία γιατί επιτρέπεται αυτό να επαναλαμβάνεται τη μια χρονιά μετά την άλλη. Αυτό είναι ντροπή για ένα ευρωπαϊκό κράτος ε, το 2017 να σταματήσετε τη συμπεριφορά αυτή. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να το χειριστούμε αυτό και θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω τους αναφέροντες που ήρθατε από τόσο μακριά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα είμαστε σε επαφή και στο μέλλον. Πρέπει να κλείσω το θέμα αυτό, διότι πρέπει να αποχωρήσω. Προτού να αποχωρήσω, θα ήθελα να καλωσορίσω θέρμα τον κύριο Μόρτεν Ράσμουσεν στο πίσω μέρος της αίθουσας που εργαζόταν για την Επιτροπή ε, αναφορών ε, πριν πολύ καιρό, μέχρι το 2004. Καλώς ήρθατε και πάλι, χαίρομαι που είσαστε εδώ πέρα. Βλέπετε, αγωνιζόμαστε ακόμα, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Ευρώπης. Ελπίζω ότι απολαμβάνετε τώρα πια την ελευθερία σας και να είστε σίγουρος ότι και εμείς ε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εγώ πρέπει να εγκαταλείψω την αίθουσα και αφήνω την Προεδρία στην Ρώσα Σαβαν Φερεκούτ και θα επανέλθω αργότερα. Θα ήθελα να Ευχαριστώ πολύ. Μου λέει η γραμματεία ότι θέλετε το λόγο, κυρία Κούνεβε, για τα λοιπά ζητήματα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που ξαναπέρνω πάλι το λόγο, αλλά ήθελα να σημειώσουμε, να μην το αφήσουμε έτσι, την πρόταση που α, οπωσδήποτε πρέπει ως Επιτροπή να κάνουμε μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια και ψήφισμα για τις συμβάσεις αυτές. Γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε πολύ αποτελεσματικά. Χωρίς την ερώτηση και το ψήφισμα νομίζω δεν το ολοκληρώσουμε καλά την διαδικασία. Ευχαριστώ. Επιμένω σε αυτό. Καλώ Καλώς. Το σημειώνουμε αλλά αφού είχε, έχουν πάρει το λόγο όλοι οι ομιλητέ και η Πρόεδρος το έκλεισε το θέμα, θα το περιλάβουμε στα πρακτικά και θα το δούμε. Δεν μπορώ να το ξανανοίξω σαν ζήτημα, αλλά το σημειώνουμε και θα το θέσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Προχωρούμε λοιπόν στο σημείο 17. Έχουμε τέσσερις αναφορές. Ναι, παρακαλώ, Ελεονόρα. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι και εγώ συμφωνώ με την κυρία Κούνεβα και τη στηρίζω. Το, θέλω να καταστήσω σαφές ότι συμφωνώ με την κυρία Κούνεβα, τη στηρίζω. Η Πρόεδρος έκλεισε το θέμα εξαιρετικά ε, νωρίς. Πρέπει να κάνουμε προφορική ερώτηση και πρόταση ψηφίσματος ως Επιτροπή. Να σημειώσετε αυτό το αίτημα και θα το συζητήσουμε στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών την επόμενη φορά η Προεδρεύουσα. Κατανοώ ότι μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης των συντονιστών. Πολλοί αναφέροντες όμως θεώρησαν ότι ε, είχε κλείσει το θέμα και έχουν φύγει και δεν μπορούμε να τους ενημερώσουμε. Αλλά το σημειώνουμε και θα το θέσουμε υπόψη της προόδου. Προχωρούμε λοιπόν στην αναφορά 0988 του 2016 Γκαμπριέλ Μοντέο για τους καθηγητές που ε, δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Πορτογαλία. 2956 επίσης αναφορά εκπροσωπεί τον Εθνικό Σύλλογο των ε, καθηγητών που εργάζονται με συμβάση ορισμένου χρόνου. Αναφορά 032 που παρουσιάζει ο Πέδρο Μαρίνιο από την Πορτογαλία για τις συνθήκες εργασίας και την αναφορά 0182, πάλι πορτογαλική αναφορά, εξ ονόματος των ε, Πορτογάλων καθηγητών. Υπάρχουν τρεις υπογραφές για ε, την αναγνώριση και επιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων. Μιλούμε για το σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης και έχει εξ ονόματος των αναφέροντων το λόγο ή δεν υπάρχουν αναφέροντες. Λοιπόν, ε, από ό,τι με ενημερώνουν, η Τζίλιαν Μουρ έχει το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να πω καταρχάς κάτι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίρνει το ζήτημα της πρόληψης της επισφαλούς εργασίας εξαιρετικά σοβαρά. Και εγώ και, ο, και οι συναδελφοί μου ε, εργαζόμαστε πολύ σκληρά στο θέμα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής οδηγίας στα διάφορα κράτη-μέλη για τα οποία ή από τα οποία λαμβάνουμε ε, προσφυγές τέτοιου είδους. Δηλαδή, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για να εφαρμοστεί η οδηγία όπως πρέπει. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση, η οδηγία βασίζεται σε μια συμφωνία πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων. Και ε, για να σας πω τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά και σε ποιο πλαίσιο εντάσσονται, θα ήταν χρήσιμο να σας πω καταρχάς με τι ασχολείται η οδηγία. Ασχολείται άμεσα με δύο ρήτρε, με δύο διατάξεις. Πρώτον, ίση μεταχείριση η ρήτρα της ίσης μεταχείρισης βασικά λέει ότι ένας εργαζόμενος που έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου θα πρέπει να την χάνει ίσης μεταχείρισης με ένα συγκρίσιμο εργαζόμενο που έχει σύμβαση αορίστου χρόνου, εκτός και αν κάτι το διαφορετικό τεκμεριώνεται επαρκώς. Δεύτερη αρχή είναι μια αρχή που ακούστηκε πολύ στην προηγούμενη συζήτηση και είναι η εξή. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να υιοθετούν μέτρα για να προλάβουν την κατάχρηση των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Αυτή η οδηγία είναι το κείμενο στο οποίο κατέληξαν οι κοινωνικοί εταίροι και θέλω να υπογραμμίσω τις παραμέτρους ε, που ε, ε, διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυστηρά και μόνο. Σε ό,τι αφορά τους Πορτογάλους αναφέροντες, Να σας δώσω ένα παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει δράση για να εφαρμόσει τα πράγματα. Ως αποτέλεσμα των σοβαρών παραπώνων και προσφυγών που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2009 μέχρι σήμερα για τη θέση των καθηγητών στην Πορτογαλία, στα πορτογαλικά σχολεία με τις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιπαραβάση κατά της Πορτογαλίας το 2010. Και Είχαμε εκτεταμένες συζητήσεις με την Πορτογαλική κυβέρνηση και στη συνέχεια μια επιστολή επίσημης κοινοποίηση, μια επιστολή τεκμηριωμένης και τηλεογημένης γνώμης που έστελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν όλων τούτου, οι πορτογαλικές αρχές ενσωμάτωσαν νομοθετικές αλλαγές στην νομοθεσία τους και αυτό σημαίνει ότι τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας πλαίσιο που είναι προσαρτημένη στην οδηγία έχουν ε, εφαρμοστεί και τηρηθεί. Ω εκ τούτου και κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό που έκαναν οι Πορτογάλοι τροποποιώντας την νομοθεσία τους που διέπει το Καθεστώ των καθηγητών δείχνει ότι η χώρα αυτή συμμορφούνται με τη Συμφωνία Πλαίσιο τη οδηγία και το 2015 για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε τη διαδικασία επί παραβάση. Αυτή την εβδομάδα μετά από συζήτηση που είχαμε με την κυρία Σοφία Ριμπέρο Ευρωβουλευτή που νομίζω ότι είναι και μέλος της Επιτροπής σας ενημερωθήκαμε ότι είναι δυνατό και πιθανό η πορτογαλική νομοθεσία να μην εφαρμόζεται στις νήσους Αζόρες για άλλους λόγους διαδικαστικούς ή νομικούς, αλλά περιμένουμε ενημέρωση σχετική. Είναι νέο ε, στοιχείο αυτό και το μάθαμε μόλις αυτή την εβδομάδα. Αυτό καταρχάς. Άρα συμπερασματικά και περιληπτικά σας λέω ότι η Επιτροπή ανέλαβε δράση, οι πορτογαλικές αρχές τροποποίησαν την νομοθεσία τους με διάφορους τρόπους, η Επιτροπή ε, εξέτασε τις αλλαγές και έκλεισε, έδωσε ένα τέλος στη διαδικασία επιπαραβάσης. Στη συνέχεια και κατόπιν τούτου έγιναν νέες πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έλεγαν ότι παραμένουν θέματα άνησης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Νέα στοιχεία δηλαδή προέκυψαν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδειχναν ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές και δεν είναι απολύτως ίση και ίδια η μεταχείριση σε ό,τι αφορά το, για παράδειγμα τις ώρες εργασίας, ε, την μισθολογική εξέλιξη και το καθεξής. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέα έρευνα για το θέμα αυτό, συνομιλώντας με τις πορτογαλικές αρχές. Έχουμε την διαδικασία διαλόγου που ονομάζουμε EU Pilot, Ευρωπαϊκή Πιλωτική Διαδικασία. Υπήρξε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πορτογαλικών Αρχών και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ε, μετά το κλείσιμο της διαδικασίας επί παραβάση ε, ερευνούμε το θέμα της άνησης μεταχείρισης. Αυτά ή ε, πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος το λόγο, μέλος της Επιτροπής μας ή κάποιος ή κάποια το λόγο. Ο Πίτερ, παρακαλώ. Φυσικά θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά με βάση αυτά που είπε η προεδρο ευχαριστω πολυ θελει κάποιο το λογο μέλο τη επιτροπης μας Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει αντιδράσει στο θέμα αυτό. Είναι θλιβερό το θέμα, αλλά κατά τα άλλα θα μπορούσε να γελάει κανείς ε, σχετικά με την επινοητικότητα των ε, κρατών μελών. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει στο θέμα. Άλλωστε είδαμε και το προηγούμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Ε, φαίνεται να είναι ένα γενικότερο πρόβλημα και κάθε κράτος μέλος προσπαθεί να δημιουργήσει τα δικά του παραθυράκια. Αλλά έχουμε ευρωπαϊκές αξίες Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Καλώς, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή πρόταση, η πρόταση του Πίτερ, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, περιμένοντας νέα στοιχεία για τις νέες προσφυγές ε, στις οποίες αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένοντας νέα στοιχεία για το τι γίνεται με τις αζόρες νήσους. Θα περιμένουμε λοιπόν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπής και Πορτογαλικών Αρχών. Περνάμε τώρα στο σημείο 18 τη ημερήσια διάταξη. Εκεί έχουμε συμπεριλάβει πέντε αναφορέ από την αυτόνομη κοινότητα τη Βαλένθια στην Ισπανία. Διάφοροι αναφέροντες θεωρούν ότι δεν εκπληρούνται τα ε, περιεχόμενα τη οδηγίας για τι συμβάσει ορισμένου χρόνου. Να δώσουμε το λόγο ευθύ αμέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι παρόντε οι αναφέροντε. Παρακαλώ. η κυρία Τζίλιαν Μουρ από την ε, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, η Ιβάνα Τρέμπ. Παρακαλώ. Thank you, Madam Um, as a... Ευχαριστώ, η κυρία Μουρ. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 και το 2013 δέχθηκε κάποιες προσφυγές που έλεγαν ότι λόγω των μέτρων που έχει θεσπίσει η αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια μειώθηκε το ωράριο εργασίας μόνο εργαζομένων ορισμένου χρόνου και άρα μειώθηκαν και οι απολαβές τους αντιστοίχως μόνο και ξεκινήσαμε βάσει του EU Pilot μία διερεύνηση ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπιστώσουμε κατά πόσο αληθεύουν οι ισχυρισμοί αυτοί και συζητήσαμε τους λόγους ε, γι' αυτό με την Ισπανική κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα αυτών των ερευνών, το EU Pilot Investigation, δείχνει ότι η αυτόνομη κοινότητα της Μπαλένθια, η δημόσια διοίκηση δηλαδή της περιφέρειας αυτή, αυτής απόσυρε το μέτρο από 1η Πρώτου του 2014. Άρα η συγκεκριμένη έρευνα για το συγκεκριμένο αυτό μέτρο έκλεισε. Και άρα θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα έχει λυθεί. Επιπροσθέτως, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των Ισπανικών ε, κρατικών αρχών σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό και τοπικό κατά πόσο εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης στον ε, δημόσιο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεχτεί και άλλες προσφυγές για διακριτική μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και υπέρ των εργαζομένων αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα, στη δημόσια διοίκηση. Και υπάρχουν με αυτή τη βάση δύο διαδικασίες επί παραβάση κατά του δημοσίου τομέα του Ισπανικού κράτους. Έχουν ανοίξει αυτές οι διαδικασίες για λόγους άνησης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου. Όμως η συγκεκριμένη αναφορά δεν είναι, ακόμα, ε, δεν είναι πια υπό εξέταση γιατί θεωρούμε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε έρθει σε επικοινωνία γραπτή με έναν από τους αναφέροντες για τα ζητήματα αυτά της Βαλένθια που αναφέρετε εσείς σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης γιατί ο αναφέρον θέλησε να ζητήσει αποζημίωση για αυτό που του είχε συμβεί στο παρελθόν. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι υπό αυτές τις συνθήκες, ε, δηλαδή ε, όταν ένα άτομο θέλει να πάρει αποσημείωση λόγω παράβασης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από πλευράς κράτους μέλους, τότε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς δεν μπορούμε να δράσουμε εξ ονόματός του. Όταν ζητά αποσημείωση πρέπει ο ίδιος να απευθυνθεί στα εθνικά δικαστήρια. Εμείς δεν μπορούμε να το πράξουμε αυτό εξ ονόματός του. Και το έχουμε υπογραμμίσει αυτό ότι μετά από τις ενδελεχείς έρευνές μας το μέτρο αποσύρθηκε, το επίμαχο και άρα σε ό,τι μας αφορά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι το ζήτημα έχει λυθεί επίσης. Η Πρόεδρος. Θέλει κάποιος το λόγο. Ο Πίτερ παρακαλώ. Ίσως θα έπρεπε στην, περί... στην περίπτωση αυτή να έχουμε την τόλμη να κλείσουμε την αναφορά. Θα ενημερωθεί ο αναφέρον Και στην περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία ανακριβή κατά τη γνώμη του αναφέροντος μπορεί να μας τα στείλει. Στην περίπτωση αυτή προτείνω να κλείσει η αναφορά, να ενημερωθεί ο αναφέρον. Εάν δεν μπορεί να δεχθεί το κλείσιμο, τότε να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Συμφωνώ να προτείνουμε. Θέλετε παρακαλώ κάτι να πείτε, κυρία Κούνεβα. Ε, προτείνω να μην κλείσει αυτή η αναφορά, γιατί το ένα θέμα έχει λυθεί, αλλά το άλλο όχι. Bueno, lo que, lo que ha dicho la Comisión. Eh... Αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι αυτές οι αναφορές έχουν λυθεί, διότι η αυτόνομη κυβέρνηση της Βαλένθια, μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά από το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση του Δικαστηρίου της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια, οι αρχές λοιπόν αποφάσισαν και αναγκάστηκαν να αλλάξουν την νομοθεσία και από 1ης πρώτου του 2014, όπως σας είπα, έχει προσαρμοστεί και υπάρχει ίση μεταχείριση στους χώρους εργασίας. Επομένως θεωρώ ότι οι αναφορές πρέπει να κλείσουν γιατί όλες έχουν λυθεί χάρη στο ανώτατο δικαστήριο της Αυτόνομης Κοινότητας της Μπαλένθια και στη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυβέρνηση της Μπαλένθια ε, οπισθοχώρησε και το έλυσε το θέμα. Τι δεν έχει λυθεί. Ε, ε, υπάρχουν νέες προσφυγές που, για άλλο θέμα που δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Επιτροπή Αναφορών. Εάν φτάσουν και όποτε φτάσουν θα τις κρατήσουμε ανοιχτές. Αυτές οι συγκεκριμένες όμως το πρόβλημά τους έχει λυθεί και γι' αυτό συμφωνώ με το Πίτερ να τις κλείσουμε, να ενημερώσουμε τους αναφέροντες και αν έχουν κάτι καινούριο να το κρατήσουμε ανοιχτές. Παρακαλώ. Ναι, αλλά το θέμα άνησης μεταχείρισης μεταξύ δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παραμένει ανοιχτό. ναι, αλλά όχι για αυτές τις αναφορές. Δεν... Δηλαδή, η αναφορά του Άγχελα Παρίθιου, του Μπερνάρντο Μπαρμπέρ, του MRR, της Κάρμεν Σάντσεθ και Θέλια Αντρές έχουν λυθεί και πρέπει αυτές τις συγκεκριμένες να τις κλείσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουμε άλλες. Άλλες αναφορές για αυτό το θέμα που θα προκύψουν στο μέλλον θα παραμείνουν βεβαίως ανοιχτές. Αλλά οι συγκεκριμένη το ζήτημά τους έχει λυθεί και θα πρέπει να τις θεωρήσουμε κλειστές και να το ενημερώσουμε τους αναφέροντες και να τις ξανανοίξουμε μόνο αν οι αναφέροντες κομίσουν, προσκομίσουν νέα στοιχεία. Εάν συμφωνείτε λοιπόν όλοι, προχωρούμε στο σημείο 19 και μιλούμε για την επίσκεψη, την ενημερωτική στη Σουηδία 21 Φεβρουαρίου και αναβλήθηκε να το δούμε αυτό στην 24-25 ε, Απριλίου 2017. Άρα, να ε, κάνουμε προτάσεις μέχρι 2 Μαΐου στις 3 Καταληκτική προθεσμία είναι 30 Μαρτίου 2017 στις 3 και ψηφοφορία 24-25 Απριλίου. Το μεταθέτουμε λοιπόν για τις 24-25 Απριλίου και καταληκτική προθεσμία 30 Μαρτίου. Ε, αν συμφωνείτε, ολοκληρώνεται η εξέταση των θεμάτων και λίγη σημερινή συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ.